Συνάδελφοι, συνεχίζουμε. Εκεί που σταματήσαμε χτες το απόγευμα, ευχαριστώ ιδιαίτερα τη Μόνικα Χολμάιερ, η οποία σήμερα το πρωί είναι εδώ μαζί μας. Θα μας παρουσιάσει τη γνωμοδότησή της για την κτηριακή πολιτική. Έχετε το λόγο, κυρία Χολμάιερ. Αγαπητέ Πρόεδρε, Ζητώ συγγνώμη που εχθές δεν μπόρεσα να είμαι εδώ, γιατί εχθές ε, μου στάλθηκαν ε, τα διάφορα έγγραφα που την Δεν μπορέσαμε δηλαδή ούτε να τα κοιτάξουμε. Έχουμε τέσσερα κτίρια, τέσσερους διαφορετικούς φακέλους. Θα προσπαθήσω να περιοριστώ στα πιο ουσιαστικά σημεία. Καταρχήν το Black Hole είναι τα κτίρια αυτό και της, το κτίριο της Μερόντ, πρόκειται για κτίρια της Επιτροπής και ουσιαστικά πτώκτηκε για ένα συμβόλαιο χρησικτησίας για 15 χρόνια, για μια χρονική περίοδο 15 χρόνια. Έχουμε επίσης το κτίριο αυτό, το πρώτο που βρίσκεται στην, ε, στο δρόμο Μοντουαγέ, πάνω από 15.000 τετραγωνικά μέτρα και το άλλο που βρίσκεται στην ε, Λεωφόρο Τερβίρεν με περισσότερα τετραγωνικά μέτρα. Είναι ένα μεγαλύτερο κτίριο. Αυτό που μας ε, αφορά εδώ είναι το θέμα της ε, των επενδύσεων αυτό, το πώς θα ενοικιαστούν αυτή την ε, έκπτωση που μας προτείνουν της τάξης του 5%. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειάζεται περισσότερα τετραγωνικά μέτρα και βεβαίως ε, εδώ έχουμε και διάφορες ε, ήδη προτάσεις για την χρήση αυτών των κτηρίων Ενδεχομένως ε, θα χρειαζόμαστε και λιγότερα τετραγωνικά από ό,τι στην αρχή είχαμε προβλέψει. Πρόκειται για τέσσερα κτίρια. Καταρχήν, για τα κτίρια αυτά έγινε μία, ένας διαγωνισμός, προκηρύχθηκε ένας διαγωνισμός. Είδαμε όμως ότι καταρχήν ε, στο Η προκήρυξη αυτή τελικά μας οδήγησε σε διάφορους συμμετέχοντες. Ο Πλάζα ήταν αυτός, η εταιρεία Πλάζα ήταν αυτή η οποία τελικά επικράτησε. Δυστυχώς δεν έχω όλα τα έγγραφα εδώ μαζί μου. Εχθές τα είχα προετοιμάσει ωραία και καλά, αλλά δεν τα βρίσκω. Λοιπόν, ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ετήσιος. Mhm. Θα επιτύχουμε σημαντικές εξοικονομήσεις στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Μιλώ για πάνω από 4 εκατομμύρια τον χρόνο και 700 80.000 για άλλα έξοδα. Και κάθε χρόνο θα έχουμε συνολικό κόστος, με συγχωρείτε μια στιγμή, ε, Λοιπόν, έλεγα ότι το ετήσιο κόστος είναι 4 εκατομμύρια 500.000 ενώ το προηγούμενο κόστος ήταν πάνω από 8 εκατομμύρια από πλευράς του ιδιοκτήτου τώρα αναλαμβάνεται και το κόστος του εξοπλισμού της τάξεως των 7 εκατομμυρίων 300.000 περίπου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν παρακαλεί τώρα να εγκριθεί ένα 8% contingency, δηλαδή ένα περιθώριο για το κόστος του εξοπλισμού, του fitting out στα αγγλικά. Εγώ προτείνω να κάνουμε κάτι που έχουμε κάνει και στο παρελθόν, δηλαδή να βάλουμε ένα 4%. Και αν ξεπεράσουν το 4% να είναι υποχρεωμένη η Επιτροπή να μας ενημερώσει. Και αυτό να το βάλουμε και στο πρακτικό αλλά και στην επιστολή προς τον Πρόεδρο. Έχω δε ενημερώσει και σχετικά τους Σκιώδη Σίγητα. Αν έχετε άλλες ερωτήσεις, πολύ ευχαρίστω να μου τις θέσετε. Αυτά είναι βέβαια για το πρώτο ακίνητο. Euh, Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν ε, ερωτήσει. Ακούσατε την εισηγήτρια για το Black Pearl και το Merod, τα δύο αυτά κτίρια της Επιτροπής. Δεν βλέπω κανέναν. Άρα αν καταλαβαίνω καλά, μέχρι 4% θα θεωρήσουμε ότι το περιθώριο είναι αποδεκτό, χωρίς παρατηρήσεις. Όταν ξεπεραστεί αυτό το 4% μέχρι το 8% θα χρειαστούν δικαιολογητικά. Και αυτό ενδεχομένως θα μπορέσει να αποτελέσει και αντικείμενο τροπολογίας για τον προϋπολογισμό του 2007, κάτι βεβαίως που θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι το τέλος Ιουνίου για να τον δούμε αυτό το προϋπολογισμό. Καθότι περιμένουμε περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τους μετανάστες και τη φιλοξενία των προσφύγων. Στις 23 Ιουνίου το βράδυ θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για όλα αυτά. Αν δεν υπάρχουν ε, όμω ερωτήσει και παρατηρήσεις, μπορούμε να ψηφίσουμε ποιο είναι υπέρ της πρόταση της εισηγήτριας. Δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε. Ωραία. Καλύτερα όμως να ψηφίσουμε. Σηκώσατε όλοι τα χέρια. Ναι. Περνάμε στην επόμενη έκθεση της κυρίας Χολμάγερ. Ακολουθεί τώρα ένα μεγαλύτερο έργο που έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πρόκειται για το τρίτο τμήμα οικοδόμησης της Καρλσρούης ε, και είναι το τρίτο μέρος που είναι και το πιο ενδιαφέρον όπως εξηγούσα. Στα προηγούμενα στάδια της κατασκευής ήταν πρώτα τα διοικητικά. Ε, υπάρχει και ε, εγκύτητα σε κάποια πυρηνικά εργαστήρια. Τα παλαιότερα είχαν μπει όλα σε ένα ενιαίο συγκρότημα. Τώρα αυτό δεν γίνεται. Τα εργαστήρια τώρα που ασχολούνται με θέματα ασφαλείας στον χώρο της ατομικής έρευνας 80% της παγκόσμιας έρευνας διεξάγεται στην Καλσρούη. Και αυτά υποτίθεται τώρα πρέπει να ε, γίνουν πραγματικά να εξυγχρονιστούν γιατί τα μηχανήματα και τα κτίρια είναι ήδη από τη δεκαετία του 70 εκεί. Άρα είναι απολύτως απαραίτητος ο εξυγχρονισμός τους. Πρώτα πρέπει να γίνει η αποδόμηση των παλαιών ε, εργαστηρίων που έχουν ε, χρησιμοποιήσει και ατομικά πυρηνικά υλικά και βεβαίως μετά να εξοπλιστούν με το πιο σύγχρονο εξοπλισμό τα νέα. Έχει γίνει μια συνεννόηση με το κρατήδιο της Βιρτεμβέργης που είναι εκεί αρμόδιο το σχετικό Υπουργείο και με το κοινό ε, ε, αυτό, ε, κέντρο ερευνών και αυτό που πρόκειται να γίνει τώρα είναι το εμβαδόν που έχουμε τώρα που είναι της τάξης των 49, των 41 μάλλον χιλιάδων ε, τετραγωνικών μέτρων. Ένα μεγάλο μέρος έως τώρα ήταν αφιερωμένο σε διοικητικούς σκοπούς. Αυτά τώρα να διαμορφωθούν εκ νέου με νέο σχεδιασμό θα χωριστούν σε διάφορα τμήματα. Ορισμένα από αυτά θα εγκαταλειφθούν μέσα στα κτίρια. Η πτέρυγα Β θα εγκαταλειφθεί μέχρι το 2035 και μάλιστα οριστικά. Η F δηλαδή μέχρι το 2025 η Γ, η G μέχρι το 2025 και μένει ακόμα ένας. Ε, ένα, μια πτέρυγα. Τέσσερις πτέρυγες λοιπόν εγκαταλείπονται. Τώρα μένει ένα μέρος το οποίο έχει το γράμμα μη και σε αυτό θα γίνονται όλες οι έρευνες στο μέλλον. Προβλέπεται η οικοδόμηση μέχρι τον Οκτώβριο 2019. Έχει γίνει η πρόσκληση εκδηλώσεως ενδιαφέροντος. Το συνολικό κόστος περίπου ανέρχεται στα 64 εκατομμύρια ευρώ. Construction works, τεχνικός εξοπλισμός, εγκαταστάσεις ασφαλείας. Επίσης ε, η, τα διάφορα τέλη και έξοδα για τους τεχνικούς εμπειρογνώμονες. Αυτά έχουν γίνει ήδη από το 2010 έως το 2015. Θα προβλέπετε και μια σχετικά μεγάλη ένα μεγάλο, ε, μεγάλο μάλλον περιθώριο τη τάξη του 20%. 20% στα αγγλικά contingency. Είναι μεγάλο το περιθώριο βέβαια, δηλαδή το περιθώριο ε, λάθους της προβλέψης, αλλά πρόκειται για εργαστήρια τα οποία χρησιμοποιούν πυρηνική τεχνολογία. Γι' αυτό και προβλέπεται, όπως εξήγησα, μια σχετικά μεγάλη contingency. Η πρότασή μου είναι, όπως πριν, από το 5% και πάνω να είναι υποχρεωμένοι να έρθουν να δικαιολογήσουν γιατί χρειάζονται περισσότερο περιθώριο. Και αυτό να περιληφθεί στην απόφαση. Συνολικό κόστος λοιπόν προβλεπόμενο τώρα είναι 64 εκατομμύρια. Από αυτά η συμβολή του ε, κοινοτικού προϋπολογισμού είναι μόνο 19%. 19% από χώρες που έχουν συμβάσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ινστιτούτο JRC που εδρεύει όπως εξήγησα στην Καρλσρούη της Γερμανίας και 62% προέρχονται από διάφορα άλλα έσοδα που επιτυγχάνει το Ινστιτούτο εργαζόμενο και διεξάγοντας έρευνες για λογαριασμό χωρών μελών. Άρα έχουμε ήδη ένα μεγάλο ποσοστό από τα 64 εκατομμύρια, δηλαδή τα 40 σχεδόν εκατομμύρια που δεν χρειάζεται να τα πάρουμε από τον κοινοτικό προπολογισμό. Εάν τώρα πάμε στο contingency, ενδέχεται να χρειαστούμε έξτρα 12 εκατομμύρια από τον κοινοτικό προπολογισμό. Αλλά όπω εξήγησα, λόγω των υψηλών απαιτήσεων ασφαλεία, κάτι τέτοιο είναι ενδεχομένω αναπόφευκτο. Αυτά πολύ σύντομα για να σα εξηγήσω ένα φάκελο που έχω λάβει από την Καρσούη, ο οποίο ήταν ιδιαίτερα ογκώδη. Μάλιστα, σα ευχαριστώ, λέει Πρόεδρο. Ευχαριστώ. Αν κατάλαβα καλά, η συμμετοχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κατά 19% σε σχέση με τον αρχικά προβλεπόμενη εκτίμηση. Το περιθώριο όμως ε, ουσιαστικά θα το αναλάβει εντελώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουν έσοδα και από τα έσοδα αυτά θα χρησιμοποιήσουν όσα παραμείνουν στα χέρια τους και στο μέλλον. Αλλά από την πλευρά του προπολογισμού δεν είναι δυνατόν να ληφθούν υπόψη αυτά τα έσοδα. Είναι ενδεχόμενα έσοδα για τα επόμενα έτη. Πρέπει λοιπόν να προβλεφθεί ήδη από τον προπολογισμό το σχετικό κονδύλι. Όπω είπα, για τα 40%. Τα δε 12, 40 μάλλον εκατομμύρια, για τα 12 εκατομμύρια από αυτά τα assigned revenues αυτοί χρησιμοποιούν ένα ε, ποσό και θα επιτύχουν έσοδα και τις επόμενες χρονιές. Όμως ακόμα δεν μπορούμε να τα βάλουμε λογιστικά μέσα στο σχεδιασμό. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Δενανό. Θα ήθελα να ξέρω κάτι παραπάνω για αυτό το πυρηνικό εργαστήριο. Τι έρευνα κάνουν, τι ακριβώς συμβαίνει, ποιες είναι οι χώρες που έχουν πρόσβαση, είναι μόνο χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και τρίτες χώρες. Μήπως θα μπορούσατε να μας παρουσιάσετε κάτι, κάποια στοιχεία για το εργαστήριο αυτό. Η συγγήτρια. Μήπως ε, για τη χρηματοδότηση μπορούσαμε να έχουμε κάποια στοιχεία. Η κυρία 28 χώρες μέλη, Ελβετία, Ουκρανία, λόγω των νέων διατάξεων του ΑΕΟ, έχει αποφασίσει λοιπόν και αυτή να συμμετάσχει. Η έρευνα αφορά αποκλειστικά ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων υφιστάμενων πυρηνικών εργοστασίων. Δεν πρόκειται για κατασκευή νέων πυρηνικών εργοστασίων. Δεν έχει καμία σχέση ε, αυτό και με την ε, πολιτική συζήτηση που διεξάγεται ούτω ή άλλω στο Κοινοβούλιο, αν θέλουμε να κατασκευαστούν νέα πυρηνικά εργοστάσια ή όχι. Πρόκειται μονάχα καθαρά για έρευνα για θέματα ασφαλεία των υφιστάμενων πυρηνικών σταθμών. Πώ μπορούν να μειωθούν οι κίνδυνοι, πώ μπορούν να βελτιστοποιηθούν οι συνθήκες ασφαλείας των υφιστάμενων ε, πυρηνικών σταθμών, διότι υπάρχουν αυτοί και λειτουργούν. Τίθεται και θέματα ε, ημιζωής, πώς θα χρησιμοποιηθούν τα διάφορα υλικά. Δηλαδή η βελτίωση της ασφάλειας υφιστάμενων πυρηνικών εγκαταστάσεων. Και όπως είπα, στο μεγαλύτερο βαθμό τους παγκοσμίως αυτές οι έρευνες διεξάγονται και στην Καλσρούη. Εντάξει, νομίζω ότι μπορούμε τώρα να τοποθετηθούμε στην έκθεση που μας παρουσίασε μόλις η κυρία Χολμάιερ. 20% είναι αυτό το περιθώριο, μέχρι το 5% δεν χρειάζονται δικαιολογητικά, πέραν το, αυτού του 5% μέχρι το 20% χρειάζεται υποστήριξη, τεκμηρίωση που θα πρέπει να υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ποιος είναι κατά? Κανείς? Είστε όλοι λοιπόν υπέρ της πρότασης αυτής. Η Στοκχόλμη τώρα και το θέμα της υγείας. Πολύ ενδιαφέρον ο φάκελος αυτός, λέει και ο το οποίο παρακολουθώ εδώ και πολλά χρόνια. Είχα κάνει κάποιες σκέψεις τότε οι οποίες δεν υλοποιήθηκαν. Ε, δυστυχώς το Σουηδικό κράτος δεν πρόσφερε υποστήριξη Επομένω, ο οργανισμός ECDC είναι η μείνει μόνο του για να αντιμετωπίσει τα θέματα. Άρα, περί τίνος πρόκειται. Πρόκειται για ένα παλαιό κτίριο το οποίο είναι χαρακτηρισμένο ως προστατευόμενο και το οποίο δεν είναι ειδώδες ό,τι αφορά τις, τους χώρους του. Απέναντι στις ανάγκες του οργανισμού ECDC. έγινε μια ε, ανάλυση αγοράς και μια πρόσκληση εκδηλώσεως ενδιαφέροντος η οποία συγκέντρωσε κάποια κτίρια. Μάλιστα στην πρώτη αυτή εκδήλωση έγινε μονάχα μια προσφορά. Στην πρώτη αυτή μάλλον πρόσκληση εκδηλώσεως ενδιαφέροντος έγινε μια μόνο προσφορά. Στη δεύτερη τέσσερις πρόσφορες όμως η περιοχή όπου βρίσκεται ε, η του οργανισμού είναι και ένα ένα σημείο της πόλης που είναι πάρα πολύ ε, ελκυστικό για πολλούς και θέλουν πολύ να εγκατασταθούν εκεί. Το μελλοντικό κτίριο, εν πάση περιπτώσει, θα έχει μεγαλύτερο εμβαδόν, δηλαδή 90.400 τετραγωνικά μέτρα. Θα διαμορφωθούν πολύ πιο αποδοτικά οι νέοι χώροι έτσι ώστε παρόλο που αυξάνει ο αριθμός του προσωπικού, αναμένεται δηλαδή για το μέλλον να αυξηθεί, παρόλα αυτά θα μπορεί στο νέο κτίριο να εγκατασταθεί καλύτερα το προσωπικό από ό,τι στο προηγούμενο. Ενώ το παλαιό είχε ανάγκη και από ανακαίνιση, που βεβαίως θα έπρεπε το κόστος αυτό να ληφθεί υπόψη Το παλαιό μίσθωμα ήταν 1,854 1.854.000. Τώρα φτάνει λίγο παραπάνω από 2 εκατομμύρια. Αλλά βεβαίω πρέπει να ληφθεί υπόψη και το κόστο τη ανακαίνιση του παλαιού, το οποίο δεν πρόκειται να δοθεί τώρα. Ο νέο ιδιοκτήτη δέχθηκε να μειώσει την προσφορά που είχε κάνει κατά 6%, κάτι που οφείλω να επικρίνω είναι το 2% τιμαριθμοποίηση. Κάποια τιμαριθμοποίηση βέβαια πρέπει να υπάρχει. Είναι κατά ο αριθμός αυτός του 2% θα προκύψει από το, την πορεία του συνολικού τιμάριθμου. Για κάθε χρόνο προβλέπεται κόστος συντήρησης της τάξης των 51.000 ευρώ. Υπάρχει και, υπάρχουν και κάποια διαρκή στοιχεία κόστους, ευνοϊκότερα όμως από ότι στο παλαιό κτίριο όπου το κόστος ανέβαινε διαρκώς και όπου ήταν ήδη 58 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Το δε fitting, out θα χρειαστεί 500.000 ευρώ, ώστε στο τέλος φτάνουμε σε ένα κόστος των 2,5 εκατομμυρίων, ενώ με το παλαιό κτίριο ήταν 2,3 εκατομμύρια, χωρίς να λεφθεί υπόψη βέβαια, όπως εξήγησα, η αναγκαία ανακαίνιση. Νομίζω ότι το νέο κόστος εν τέλει αποτελεί και την οικονομικότερη λύση, διότι δεν προκύπτει πλέον κόστος ανακαίνισης. Σας ευχαριστώ για την ε, σαφήνεια των προτεσιών σας. Υπάρχουν παρατηρήσεις ή ερωτήσεις. Δεν βλέπω. Μπορώ λοιπόν να θεωρήσω ότι η Επιτροπή Προϋπολογισμών δεν αποδοτεί θετικά σε αυτό το σχέδιο για το εισήντηση e στη Στοχόλμη. Ωραία, ευχαριστούμε. Κύριε Χολμάιερ για το ΕΑΣΟ. Θέλετε, από ό,τι κατάλαβα, δύο τις εβδομάδες για να γνωμοδοτήσετε. Ε, κυρία θα ήθελα να προτείνω, κύριε Πρόεδρε, να κάνουμε κάτι άλλο. Όπως κάνει και το Συμβούλιο δηλαδή. Αυτά που έχει δώσει τώρα η ΕΑΣΟ είναι ένα είδος προπληροφόρησης, ένα pre-warning το αποκαλούν μάλιστα. Εγώ είμαι απολύτως ανοιχτή στο θέμα αυτό, διότι η ΕΑΣΟ είναι ήδη κατεστημένη στα κτίρια. Γνωρίζει καλά τα κτίρια, γνωρίζει ότι χρειάζεται επέκταση των κτιρίων. Θα έπρεπε αυτό το pre-warning να έχει γίνει νωρίτερα. Ακόμα διαρωτώ πόσα γραφεία αποκτούμε περισσότερα στην περίπτωση αυτή. Λένε για internal area και external area δεν μας λένε ούτε εκατοστό. Γι' αυτό λέω ότι σε δύο εβδομάδες, εγώ καταρχήν είμαι υπέρ, διότι όντως η ΕΑΣΟ θα χρειαστεί χώρους και έχουν όντως οικοδομηθεί οι χώροι αυτοί. Να θυμόμαστε όμως ότι ο οργανισμός αυτός ήταν κάτι το οποίο το θέλαμε οπωσδήποτε. Αν θέλουν τώρα να διαπραγματευτούν τιμές μαζί μας που δεν πληρώνουμε ούτε καν, δεν καταβάλουμε ούτε καν για το κέντρο των Βρυξελών, ε, τότε στέκομαι κάπως επικριτικά απέναντι στο ενδεχόμενο αυτό. Διότι θα πρέπει εν, τέλος, ε, θα πρέπει εν τέλει μάλλον και η Μάλτα, γιατί εκεί είναι, εκεί, γι' αυτό το κράτος μιλούμε, θα πρέπει να δείξει κάποια ευκαμψία, διότι και άλλες χώρες είχαν δείξει έντονο ενδιαφέρον να αποκτήσουν την έδρα του εν λόγω οργανισμού. Άρα, να προχωρήσουμε, αλλά όχι στην τιμή των 250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Νομίζω λοιπόν ε, να κάνουμε μια προσπάθεια να κατεβάσουμε τις τιμές αυτές. Νομίζω ότι έχει μεν νόημα το έργο αυτό, αλλά να δούμε και αυτή την, προ... την ε, προειδοποίηση γιατί η υπογραφή πρόκειται να μπει το αργότερο σε τέσσερις εβδομάδες, διότι πρέπει να φύγουν από το κτίριο, από το παλαιό κτίριο. Στο νέο κτίριο είναι εγκατεστημένε κάποιες υπηρεσίες του Μαλτέζικου Δημοσίου και οφείλουν να αποχωρήσουν. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε τι 24 Ιουνίου, δεδομένου ότι μπορούμε να δούμε το θέμα πριν από τι 24 Ιουνίου. Ευχαριστούμε. Εάν μα στείλουν το ερωτηματολόγιο να γνωρίζουμε περί τίνος πρόκειται και τι θα ψηφίσουμε και να γνωρίζω και εγώ να μπορώ να σας πω δηλαδή τι ακριβώ καλούμαστε να πληρώσουμε διότι δεν ξέρουμε ακριβώς τα νούμερα. Μένουμε εκτεθειμένες στην περίπτωση αυτή και το ίδιο βεβαίω και ο οργανισμό ΕΑΣΟ. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώνεται λοιπόν αυτό το ζήτημα για τα κτίρια. Έτσι λοιπόν θα μπορέσουμε να περάσουμε στο διορθωτικό προϋπολογισμό υπαριθμών 2 του 2016. Ah non, Όχι, με συγχωρείτε. Θα ξεκινήσουμε από την Ιορδανία και το Λίβανο. plusieurs d'entre nous. εξημών. Θα βγήκαμε σε αποστολή στη Μέση Ανατολή από τις 16 ε, έως τις 19 Μαΐου και επισκεφθήκαμε διαδοχικά την Ιορδανία και το Λίβανο. Συναντήσαμε τις τοπικές αρχές, τις εθνικές αρχές, τις περιφερειακές αρχές, και συναντήσαμε ε, διάφορους που είναι επιτόπου, είτε Επιτροπή Προσφύγων, που ανήκει στον ΟΗΕ, είτε πρόκειται για την Ίνρα, τον οργανισμό που δημιουργήθηκε το 1948 και προσφέρει αρρωγή στους ε, Παλαιστίνιους πρόσφυγες ή σε όσους βρίσκονται στην περιοχή. Επίσης, συναντηθήκαμε με μη κυβερνητικέ οργανώσεις και φυσικά με πρόσφυγες. Μεταβήκαμε σε καταβλισμούς, σε αναγνωρισμένους επίσημα καταβλισμούς, όπως στην Ιορδανία, όπου έχουμε τρεις καταβλισμούς. Και πήγαμε στον καταβλισμό της ΑΣΡΑΚ, όπως σήμερα εκεί φιλοξενούνται περίπου 50.000 άτομα στη μέση της ερήμου και φυσικά όταν ε, ήμασταν εκεί ήταν 42 βαθμοί η θερμοκρασία και ε, μπορείτε να φανταστείτε ε, τη θερμοκρασία που έκανα μέσα σε αυτά τα κτίρια. Επίσης, όπως σας είπα, υπάρχουν τρεις καταβλισμοί στην Ιορδανία, αλλά εκεί δεν χωρούν μόνο το 20% παρά μόνο το 20% των σύρων προσφύγων. Το ίδιο και στην Τουρκία. Σε ό,τι αφορά το Λίβανο, δεν υπάρχει αναγνωρισμένος επίσημα καταβλισμό. Ε, υπάρχουν ουσιαστικά κάποιο κατασκηνώσεις, ε, κατασκηνώσεων, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, και μπορούμε να πούμε ότι οι συνθήκες ε, είναι κάπως επισφαλεί. και δυστυχώς αυτό δεν τιμά την κατάσταση. Έχουν κατασκευαστεί σκηνέ με κάποια ανακυκλωμένα υλικά και πληρώνεται ενίκιο για τη γη όπου βρίσκονται και φτάνουμε στο ενίκιο στο 90, 100 δολάρια ως 100 δολάρια το μήνα και φυσικά περίπου πληρώνεται και ίδιο ποσό για το ρεύμα. Εκεί Συναντάμε συνήθω οικογένειε, γυναίκες και πολύ μικρά παιδιά, γιατί συνήθω οι άντρε δουλεύουν παράνομα και καθώς δεν έχουν πόρους οι άνθρωποι αυτοί, η εξωτερική όρη είναι 12 δολάρια τη μέρα για ένα υλικό και 4 δολάρια για ένα παιδί. Και σε αυτές τις συνθήκες ε, επιλέγουν οι οικογένειες να το παιδιά τους να εργαστούν παρά στο σχολείο. Πρόκειται λοιπόν ε, για ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Συνολικά, στο Λίβανο έχουμε 1.700.000 ε, πρόσφυγες από τη Συρία σε ένα πληθυσμό 6 εκατομμυρίων κατοίκων και στην Ιορδανία 650.000 Σύρους πρόσφυγες, ίσως και περισσότερους. Ε, εμείς στο ΑΣΡΑΚ, στον καταβλισμό, που επισκεφτήκαμε, που βρίσκεται στην βορειοανατολική Ιορδανία. Στους 50.000 προστίθενται 200-300 νεοφυχθέντες. Καθημερινά είναι κλειστά τα σύνορα και μάλιστα μιλάμε για τα βορειοανατολικά. Ο πρόεδρο Ομπάμα σε πρόσφατη επίσκεψη ξεπίεσε στι Ιορδανικέ Αρχέ και μπόρεσε να πετύχει μια συμφωνία συμπληρωματική υποδοχή περίπου 20.000 ατόμων και αυτοί με το σταγονόμετρο γίνονται δεκτοί, 200-300 την ημέρα και από την πλευρά της Συρίας, τα Συριακά σύνορα περιμένουν άνθρωποι σε ιδιαίτερα καταστροφικές συνθήκες από ανθρωπιστική σκοπιά. Πρόκειται για συνθήκες πραγματικά άθλιες. Και επίσης συναντήσαμε πρόσφυγες εκτός των καταβλισμών. Σκέφτομαι το πράστιο Λαμάνο που εκεί επίσης είδαμε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες σε προσωπικό επίπεδο, πολύ δύσκολες καταστάσεις, ανθρώπους που είναι παράνομοι, προδήλως και οι αρχές μπορούν να ασκήσουν διάφορες πιέσεις επάνω τους αλλά οι ανθρωπιστικές οργανώσεις και οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις είναι παρούσες εκεί και χάρη σε αυτές μπορέσαμε να κάνουμε αυτή τη διαπίστωση. Πρέπει να παρατηρήσουμε το εξής, ότι η υποδοχή των προσφύγων είναι μία από τις ε, όψεις της κρίσης που πλήττουν όλη την περιοχή. Η οικονομία υποφέρει, καθώς είναι κλειστά τα σύνορα, είναι περιορισμένες οι αγορές και στις συνθήκες αυτές υπάρχει και η αβεβαιότητα του πολέμου. Δυστυχώς ε, η πραγματικότητα στη Συρία είναι δραματική. Χτες μάλιστα είχαμε ένα νέο δράμα. Έτσι λοιπόν οι επενδύσεις, οι παραγωγικές επενδύσεις που προέρχονται από ξένους επενδυτές δεν φτάνουν εκεί. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να πυροδοτεί μια λυσίδα γεγονότων που πλήττουν τα συμφέροντα. Έτσι λοιπόν, καθώς δεν υπάρχει ανάπτυξη και επενδύσεις, είναι υψηλή η ενεργεία και βρισκόμαστε σε ένα είδος εντάσεων που υπάρχει μεταξύ των ντόπιων και των προσφύγων γιατί νιώθουν ότι τους ανταγωνίζονται οι πρόσφυγες. Και αισθανόμαστε αυτή την ένταση. Συναντήσαμε στη Βρυτό, στο Λίβανο, βουλευτές και είδαμε ότι υπάρχει έλλειψη κατανόηση από τις τοπικές αρχές. Παραδείγματο χάρη, μια μητέρα απευθυνθήκε στον Υπουργό Εσωτερικών στο Λίβανο και ζήτησε χρήματα για να ε, μπορέσει να κάνει κάποιες εργασίες ε, στο σχολείο και της είπε υπουργός ε, αν έχεις παιδιά πρόσφυγες μπορούμε να σε βοηθήσουμε αλλά αν δεν έχεις παιδιά προσφύγων δεν υπάρχουν χρήματα. Αισθανόμαστε λοιπόν πως διαμορφώνεται αυτή η τεταμένη κατάσταση και όλη βοήθεια που μπορούμε να δώσουμε στους πρόσφυγες είναι πολύ μικρή και υπάρχει και πληθυσμός κάτω από το κατόφλι από το της φτώχειας και στην Ιορδανία και στο Λίβανο και μερικές ε, φορές ε, οι ντόπιοι μπορούν να βλέπουν και με κάποιο φθόνο αυτά που δίνονται στους πρόσφυγες. Ε, μπορώ να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ σύντομα απάντησε πολύ γρήγορα απάντησε στις δραματικές συνθήκες που πλήγουν τη Συρία μέσω του Κατεπιστευτικού Ταμείου για τη Συρία, το Ταμείο Μαντάντ, το οποίο δημιουργήθηκε το Δεκέμβριο του 2014 και από το 2011 μπορούμε να πούμε ότι μέσω των πιστώσεων ε, του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά στην Ιορδανία έχει τετραπλασιάσει τη βοήθειά της πρακτικά. Έχει διπλασιάσει τη ο Πρόεδρος. Έχει συνεισφέρει 1,3 δις και στο Λίβανο έχουμε τετραπλασιάσει τη βοήθεια και φτάσαμε στα 980 εκατομμύρια. Και αυτό χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη την ανακοίνωση που έγινε στην έκβαση της Συνόδου στο Λονδίνο το Φεβρουάριο και προσθέσαμε εκεί μια δέσμευση ενός επιπλέον δισεκατομμυρίου. Αυτό μας επέτρεψε να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε αυτό που εννοούσαμε με την έννοια του συμπαγούς. Αυτό ορίστηκε στην Σύνοδο του Λονδίνου ε, πρόκειται για μια σύμβαση που συνδέει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις υπογράφουσες χώρες που πρέπει να αναλάβουν δεσμεύσεις σε ό,τι αφορά θεμελιώδεις απαιτήσει, είτε μιλάμε για άδειες παραμονής, οι άδειες παραμονής στο Λίβανο κοστίζουν 200 δολάρια ανά άτομο, άνω των 14 ετών Δηλαδή, αν ε, έχουμε παράνομους προσφύγει, φυσικά δεν μπορούν να πληρώνουν ετησίως 200 δολάρια και η άδεια εργασία Η Ορδανία προχωρά σε μια διαδικασία για να ευνοήσει την απασχόληση των προσφύγων. Σήμερα απασχολεί περίπου 500.000 Αιγυπτίους και αν μπουν και πρόσφυγες στην αγορά εργασίας, από ό,τι φαίνεται θα πρέπει κάποιοι Αιγύπτιοι να επιστρέψουν στην χώρα προέλευσής τους. Και έτσι λοιπόν μπορούμε να μετακινήσουμε τις δυσκολίες και από ό,τι φαίνεται 500.000 Ιορδανοί μεταξύ αυτών που έχουν τη μεγαλύτερη ευχέρεια να έχουν εκπαίδευση εργάζονται σήμερα στις χώρες του κόλπου. Αλλά είναι κάπως διαφορετική η κατάσταση στις χώρες του κόλπου. Έχει αλλάξει λόγω της εξέλιξης των τιμών στο πετρέλαιο και των ορυκτών καυσίμων. Έτσι λοιπόν δεν είναι σταθερή η κατάσταση. Τι διαπιστώσαμε λοιπόν. Ότι στην ε, υπάρχει μία κυβερνητική εξουσία λαμβάνει η κυβέρνηση αποφάσει και τι κάνει σεβαστές. Αντίθετα στο Λίβανο δεν υπάρχει παρουσία τη δημοκρατίας εδώ και δύο χρόνια και οι κυβερνητικέ οργανώσεις είναι ιδιαίτερα πολύπλοκε. Πήγαμε στην κοιλάδα τη Μπεκά και εκεί συναντήσαμε κάποιους ανθρώπους, ένα δήμαρχο που μας είπε μην ασχολείστε με την κυβέρνηση, μην χάνετε το χρόνο σας. Αν θέλετε να κάνετε συγκεκριμένα πράγματα, εδώ πρέπει να επικεντρωθείτε και όχι σε κυβερνητικό επίπεδο. Συναντήσαμε επίσης ε, και κάποιον ε, αρμόδιο που ασχολείται στον τομέα του νερού και επισκεφτήκαμε ένα κέντρο ε, που ε, αφορά την επεξεργασία των λιμάτων ε, και ένα άλλο κέντρο για την επεξεργασία του πόσιμου νερού και τα δύο αυτά λαμβάνουν βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να λειτουργήσουν. Συμβαίνουν λοιπόν ενδιαφέροντα πράγματα εκεί. Ακούσαμε και υπουργού, ιδίω στο Λίβανο, να μας λένε ότι θα μπορούσαμε να τα κάνουμε όπως οι Τούρκοι και να επιτρέψουμε στους πρόσφυγες ε, να ακολουθήσουν τη θαλάσσια εδώ για να πάνε στην Ευρώπη. Σκεφτείτε ε, <laughs> ουσιαστικά το εκατομμύριο που έχουμε εκεί με σύγκριση, σύγκριση με τα έξι δισεκατομμύρια που έχουμε δώσει στην Τουρκία. Αυτό που μας εξέπληξε είναι οι συνθήκες ε, της ε, εκπαίδευσης για τους νέους. Το ίμιση των νέων που προέρχονται από αυτές τις οικογένειες των προσφύγων δεν πηγαίνουν στο σχολείο. Όταν ε, μιλάμε για ένα-δύο μήνες, ίσως να μην είναι πολύ σοβαρό, αλλά εδώ μιλάμε για χαμένες γενιές. Υπάρχει τέτοιο κίνδυνος. Και στους καταβλισμούς που επισκεφθήκαμε, στο ΣΡΑΚ, οργανώνουμε το σχολείο, ε, σε δύο βάρδιες από τις 7 στο μεσημέρι και η δεύτερη βάρδια είναι από τις 12 μέχρι τις 5 το απόγευμα σε δύσκολες συνθήκες, κάνει πολύ ζέστη και δεν ξέρω τι σκεφτονται οι συνάδελφοι αλλά έχω μια ανάμνηση πολύ σημαντική συναντήθηκα με ένα νέο 17 ετών και είχε πάει για κάποιες ώρες ε, μόνο στο σχολείο και προσπαθήσαμε να τον προετοιμάσουμε να περάσει το διαγωνισμό για να πάει στην ανώτατη εκπαίδευση. Και μας ρώτησαν οι νέοι αυτοί <laughs> ποιο είναι το μέλλον μας. Εγώ θυμάμαι πραγματικά το βλέμμα τους ήταν πάρα πολύ σοβαρό. Καλώς συνειδητοποιούσαν ότι η ζωή τους, το μέλλον τους ίσως ήταν ανύπαρκτο και μπορούμε να φανταστούμε τις συνέπειες σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και ποια οδό θα μπορούσαν να πάρουν αυτοί οι νέοι σε αυτές τις συνθήκες, ποια πορεία θα μπορούσαν να ακολουθήσουν. Και ε, Ξέρετε, ε, όταν μιλάμε για ε, τις συνθήκες, ε, παραδείγματος χάρη δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα. Επίσης, επισκεφτήκαμε σχολεία, ένα σχολείο της UNICEF στην Ιορδανία και στο Λίβανο. Είδαμε εκεί πολύ ισχυρή δέσμευση από τους εκπαιδευτικούς για να βρουν τα κονδύλια, πρέπει να κατασκευαστούν σχολεία. Όμως αυτή τη στιγμή έχουμε όπως σας είπα δύο βάρδιες από τις 7 στις 12 και από τις 12 στις 5 το απόγευμα. Ακούσαμε γονείς που μας είπαν πώς εκτιμούν τις ε, συνθήκες ε, στις οποίες πηγαίνουν τα παιδιά σχολείο. Βέβαια, ό,τι έχουμε πετύχει πρέπει να αναγνωριστούν και να ενθαρρυνθούν. Επίσης, επισκεφθήκαμε κοινωνικά κέντρα που λειτουργούν ως ε, κλινικές και κέντρα φροντίδας και είδαμε πως η πατερμοστία το Ηνωμένων Εθνών για τις Πρόσφυγες ε, απευθύνει έκκληση σε θελοντές που επιλέγονται μεταξύ των προσφύγων. Ένας θελοντής για χίλιους πρόσφυγες είναι επιτόπου, βλέπουν ποιε είναι οι ανάγκες του πληθυσμού, ακούνε τον πληθυσμό για να δώσουν συμβουλές, παίρνουν το σχάρι σε κάποια γυναίκα, να την παραπέψουν ε, σε ένα κέντρο συμβουλών ιατρικών επίσης για τα θέματα των σχολείων. Ε, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μπορεί να είναι πάρα πολύ μακριά από τα σχολικά κτίρια. Έτσι λοιπόν τίθεται και το θέμα πώς θα μαζέψουμε αυτούς τους ανθρώπους για να πάνε στο σχολείο. Και θα πρέπει να οργανώσουμε και συστήματα συλλογής των ανθρώπων αυτών. Συγκέντρωσής τους για να πάνε στο σχολείο. Είπατε η αρμοστία τους ε, δίνει 170 δολάρια το μήνα και αυτό προκαλεί κάποια ερωτηματικά γιατί μπορεί να παίρνουν ε, τα επιδόματα αυτά κάποιοι άνθρωποι που δουλεύουν στην ε, παραοικονομία και κάποιοι πιστεύουν ότι τελικά αυτά τα επιδόματα μπορεί να μην τους ενθαρρύνουν να εργαστούν. Υπάρχει μια εσωτερική συζήτηση ε, κάπως ε, μπερδεμένη εδώ και να σας πω ότι εγώ κρατάω δύο διδάγματα, δύο συστάσεις που με εμπνέουν. Αυτά βασίζονται στην αρχή της αμοιβές εμπιστοσύνης Δίχως αυτή νομίζω ότι κάθε συνεργασία είναι μάταιη. Καταρχήν πρέπει να πετύσουμε από τις αρχές της Ιορδανίας και του Λιβάνου την μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια και να μας παρέχουν δημοσιονομικά και οικονομικά έγγραφα. Οι βουλευτές, οι Λιβανέζοι, με τους οποίους συναντηθήκαμε, μου προκάλεσαν κάποιες αμφιβολίες σας είπα σε ποιες συνθήκες ε, λειτουργεί η κυβέρνηση. Σίγουρα μπορεί να υπάρχει πρόοδο σε ό,τι αφορά τα δημοσιοοικονομικά του Λιβάνου. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι σαφής. Θα πρέπει να πετήσουμε ως αντάλλαγμα της βοήθειάς μας από τους εταίρους μας κάποιες ελάχιστες αρχές. Όμως, η δεύτερη σύστασή μου είναι η εξής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως αντάλλαγμα δεν θα πρέπει να είναι πλέον ιστερική σε ό,τι αφορά το γραφειοκρατικό ζήτημα. Έχουμε τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες. Είναι πάρα πολλοί. Είναι πολύ άριθμοι λοιπόν εκεί. Αλλά ουσιαστικά ο Ίνρα αποτελεί κράτος εν κράτη. Έχει συσταθεί από τα Ηνωμένα Έθνη για να βοηθήσει τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες. Και υπάρχουν λοιπόν παλαιστίνικες κοινότητες επιτόπου, αναγνωρίζοντας τέτοιες. Και υπάρχουν και σχολεία του Ίνρα, υπάρχουν κοινωνικά κέντρα του Ίνρα, υπάρχουν ε, κλινικές και ο προϋπολογισμός του Ίνρα ουσιαστικά είναι κατά κάποιο τρόπο ο κρατικός προϋπολογισμός που συμμετέχει στην παροχή αλληλεγγύης στους Παλαιστίνους πρόσφυγες αν χρειάζεται ε, ίνρα εδώ ε, και ευρωπαϊκές φωνές, εμείς εδώ μπορούμε να υπερασπίσουμε την, ε, τον ίνρα. Υπάρχει παρουσία και στη Λωρίδα της Γάζας και σε όλες τις γειτονικές χώρες του οργανισμού αυτού. Για το 2015 η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη διοργάνωσε δέκα διαφορετικούς ελέγχους από τις διάφορες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η UNICEF θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ των διαφόρων που συνεισφέρουν είναι ο οργανισμός που απαιτεί την μεγαλύτερη τεκμηρίωση με εξάντε ελέγχους, με δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλονται με πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Αυτό όπως ακούγεται πολλές φορές, δημιουργεί θέσεις απασχόλησης. Και όλοι οι υπεύθυνοι που συναντήσαμε επί τόπου μας εξήγησαν ότι αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν ενδεχομένως να χρησιμοποιούνται με πιο χρήσιμο τρόπο αν δεν διοχετευόταν σε γραφειοκρατικές διαδικασίες, αλλά θα μπορούσαν να είναι πολύ πιο ε, χρήσιμα για την πραγματική ανθρωπιστική βοήθεια. Μας είπαν μάλιστα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πολλές φορές δαπανά στη γραφειοκρατία ένα τμήμα των κονδυλίων. Σήμερα το πρωί ήμουν στην παρουσία της κυρίας Καλβίνιο που μιλούσε για την αποτελεσματικότητα της Ευρώπης και μίλησα ακριβώς για αυτή την αποστολή μας και ε, για όλα αυτά που είδαμε στην Ιορδανία και στο Λίβανο. Η αποτελεσματικότητα λοιπόν σίγουρα προϋποθέτει πιο αποτελεσματική χρήση και βεβαίως εκ των υστέρων ελέγχους και απόδοση λογαριασμών με μεγάλη ακρίβεια. Εμείς σαν Επιτροπή Προϋπολογισμού θα πρέπει να μπορούμε όταν κάνουμε τέτοιου είδους ταξίδια να έχουμε απλά έγγραφα, σαφή έγγραφα τα οποία μας δείχνουν όλες τις ροές τι ήταν η δέσμευση, τι τελικά πραγματοποιήθηκε και ποια είναι τα πραγματικά κονδύλια που είχαν δεσμευθεί και που χρησιμοποιήθηκαν. Δεν είδαμε τέτοιου είδους έγγραφα. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσουν εδώ μαζί, μας, μαζί μου και οι συνάδελφοι. Ακούσαμε πολλά λόγια, διαβάσαμε πολλά, αλλά τελικά δεν είδαμε συγκεκριμένα έγγραφα όσον αφορά την απόδοση των λογαριασμών. Και είμαστε η Επιτροπή Προϋπολογισμού. Αυτά. Είχα να πω για αυτή την αποστολή και το λέω εξ ονόματος όλων των συναδέλφων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τις δύο αντιπροσωπείες που μας υποδέχθηκαν της Ευρωπαϊκής Ένωσης μία στην Ιορδανία, αλλά και στο Λίβανο, οι οποίοι οργάνωσαν συναντήσεις με όλους τους ε, δωρητές, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τα Ταμεία Ανάπτυξης, ε, εδώ μιλάω για γαλλικούς φορείς, αλλά και άλλοι γερμανικοί οργανισμοί. Σίγουρα χρειάζεται καλύτερο συντονισμό γιατί υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν όμως και κάποιες διμερείς σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών και των φορέων επιτόπου. Είχαμε μαζί μας και την ε, πρόεδρο της αντιπροσωπείας, την κυρία Ματίας, Ευρωπαϊκή Ένωση Χώρες του Μασρέκ, η οποία μας βοήθησε με την εμπειρία της και τη γνώση της. Ευχαριστώ ιδιαίτερα και την γραμματεία της Επιτροπής Προεπολισμού, τον Κιγιόμ Μρέι και όλους τους συνεργάτες για την πολύτιμη στήριξή τους. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον ταξίδι με φορτωμένο πρόγραμμα και θα ήθελα να πω ότι ίσως θα ήταν χρήσιμο να περνάμε λίγο περισσότερο χρόνο επί τόπου. Και επαναλαμβάνω, όταν ψηφίζουμε ένα προϋπολογισμό, βλέπουμε τα νούμερα, βλέπουμε τις δεσμεύσεις, Πολλές φορές όμως δεν βλέπουμε στην πράξη πώς χρησιμοποιούνται αυτά τα κονδύλια. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για τις χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας. Βεβαίως εγώ ανέφερα τα προσωπικά μου σχόλια και φυσικά θα συμπληρώσετε. Ευχαριστώ. Εσείς κάνατε μια πρώτη παρουσίαση των όσων ζήσαμε και είδαμε σε αυτή την αποστολή, αλλά θα ήθελα και εγώ καταρχήν να ξεκινήσω με τις ευχαριστίες, γιατί είναι αλήθεια ότι η Γραμματεία προετοίμασε μια πλήρη αποστολή με πολύ βεβαρημένη ατζέντα, αλλά μπορέσαμε να δούμε τόπου τα σχέδια που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μπορούσαμε να έχουμε και συνεδριάσεις με διάφορους διεθνείς οργανισμούς που εργάζονται εκεί και μπορέσαμε να συναντηθούμε και με εκπροσώπους των κυβερνήσεων. Ήταν ισορροπημένη λοιπόν η ατζέντα και φυσικά υποστηρίχθηκε η δουλειά της ε, γραμματείας από τις δύο αντιπροσωπείες που έχουμε στο ΜΑΝ και στη Βρυτό. Κάνουν φανταστική δουλειά επί τόπου και ήταν πάρα πολύ χρήσιμες όλες οι πληροφορίες που μας παρήχαν. Είναι αλήθεια ότι δεν έλειπαν πληροφορίε. Πολλέ φορέ είχαμε πάρα πολλέ πληροφορίε και πολλά αριθμητικά στοιχεία και ίσω μα κόστησε λίγο να σχηματίσουμε την πραγματική εικόνα, αλλά όχι λόγω έλλειψη πληροφοριών, ακριβώ λόγω του αντιθέτου. Αυτέ οι αποστολέ είναι πάρα πολύ σημαντικέ. Γιατί όταν εδώ συζητούμε τις τροπολογίες και βλέπουμε αν μπορούμε να βρούμε ένα περιθώριο για να μπορέσουμε να βάλουμε ακόμα ένα εκατομμύριο ε, Παραδείγματο χάρη συμβαίνει συνήθω σε αυτή την επιτροπή μια τέτοια συζήτηση. Ακόμη και αν ξέρουμε τι υπάρχει ε, από πίσω, δεν το έχουμε αισθανθεί. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικέ αυτέ οι υποστολέ εκεί επί τόπου. Με τι επόμενε διαπραγματεύσει νομίζω ότι θα είναι πολύ πιο εύκολο να φτάσουμε σε συμφωνίε, γιατί είδαμε πόση διαφορά κάνουν τα χρήματα που διαπραγματευόμαστε εδώ και στη συνέχεια με το Συμβούλιο. Μπορούσαμε να, να δούμε τις συνθήκες στις οποίες ζουν οι πρόσφυγες στην Ιορδανία και στο Λίβανο και επίσης ε, βλέπουμε ότι και τα χρήματα μας επιτρέπουν να χρηματοδοτήσουμε σχολεία, νοσοκομεία, επεξεργασία, κέντρο επεξεργασία λιμάτων ή νερού. Δεν αρκούν όλα αυτά, αλλά τουλάχιστον είναι μια μεγάλη βοήθεια. Και ακόμη και αν οι πρόσφυγες αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε ιδιαίτερα επισφαλείς συνθήκες. Δεν ξέρω τι θα είχαν απογίνει αν ούτε καν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έκανε αυτή την οικονομική προσπάθεια για να τους βοηθήσει. Και νομίζω ότι γι' αυτό πρέπει να συνεχίσουμε την παροχή υποστήριξης δημοσιονομικά στις χώρες αυτές. Όπως σας είπα, όχι μόνο στους πρόσφυγες, αυτό ήταν ένα μήνυμα που προσπαθήσαν να στείλουν και την προσωπία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι μόνο λοιπόν στήριξη στου πρόσφυγε, αλλά είναι υποστήριξη σε όλα τα ευάλωτα άτομα που ζουν στο Λίβανο και στην Ιορδανία. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφοροποίησει. Αυτοί που χρειάζονται τη βοήθειά μα θα τη λάβουν ανεξάρτητα από την προέλευσή του, τη θρησκεία του και το φύλλο. Νομίζω ότι πρέπει να συνειδητοποιούμε ότι το μέλλον των ανθρώπων αυτών είναι ιδιαίτερα βέβαιο. Και όταν συναντήσαμε αυτά τα παιδιά, τα 17χρονα, είδαμε το βλέμμα τους που έλεγε «Τι κάνω εδώ, σημαίνει κάτι, χρησιμεύει σε κάτι, το ότι σπουδάζω, θα μπορέσω κάποια στιγμή να επιστρέψω στη χώρα μου, να πάω σε ένα πανεπιστήμιο». Πράγματι ήταν πολύ σκληρή αυτή η συνάντηση. Και όχι μόνο με αυτά τα παιδιά, ζήσαμε και στιγμές ε, με οικογένειες που έχουν ε, παιδιά με πάρα πολλά σωματικά και ψυχικά προβλήματα και μας ρωτούσαν τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να λύσει τις αιτίε όλων αυτών, γιατί εμείς δίνουμε ε, βασική βοήθεια, αλλά αν δεν λύσουμε το τι συμβαίνει στη Συρία, απλώς ε, βάζουμε έναν επίδεσμο. Αλλά φυσικά μπορούσαμε να επισκεφτούμε και σχολεία και είδαμε τα παιδιά να χαμογελούν και νομίζω ότι η δουλειά που γίνεται κυρίως στο Λίβανο δηλαδή να έχουν πρόσβαση τα παιδιά στην εκπαίδευση. Μας ε, διαβεβαίωσαν ότι 450.000 παιδιά που είναι πρόσφυγες αυτή τη στιγμή, από αυτά 200.000 πηγαίνουν στο σχολείο και το Σεπτέμβριο θα μπορέσουν να στείλουν στο σχολείο και τα 450.000 παιδιά. Είναι τεράστια αυτή η προσπάθεια ε, φανταστείτε αν το μεταφέραμε αυτή την προσπάθεια εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να συνεχίσουμε να του υποστηρίζουμε. Επίση είναι πολύ επισφαλεί οι συνθήκε διαβίωσή του. Φυσικά όλα μπορούν να βελτιωθούν, μπορούμε να πετύσουμε πολλά περισσότερα από τι κυβερνήσει τη Ιορδανία και του Λιβάνου ή από τη μη κυβέρνηση του Λιβάνου στην περίπτωση αυτή, αλλά τέλο πάντων ο Υπουργό Παιδεία ε, κάνει φανταστική δουλειά αυτή τη στιγμή. Επίσης, ε, εμείς με τη δική μας πολιτική δεν μπορούμε να κάνουμε να δίνουμε και μαθήματα, ούτε είμαστε παράδειγμα. Πρέπει λοιπόν να το αναγνωρίσουμε αυτό και να βοηθήσουμε αυτές τις δύο χώρες έτσι ώστε να μπορούν να δώσουν κάποιο νόημα στη ζωή των προσφύγων και των Συρών αλλά και των Παλαιστίνιων που είναι μεγάλη πλειοψηφία. Ένα μόνο στοιχείο. Ο Λίβανος με τον πληθυσμό των 4 εκατομμυρίων γιατί έχει ε, και 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγε περίπου έχει δεχτεί πολύ περισσότερου πρόσφυγε από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό λοιπόν αξίζει να το στηρίξουμε. Oui. Ε, κύριε Ομαρζή. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για αυτή την παρουσίαση που μας κάνατε δεν είναι εύκολο. Είναι ρεψοκίνδυνο θα έλεγα μάλιστα γιατί πρόκειται για περίπλοκες ε, καταστάσεις αυτές που συναντήσαμε στην Ιορδανία και στο Λίβανο. Πρόκειται για έντονες καταστάσεις καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της ε, επίσκεψης. Όσον αφορά τις δικές μου εντυπώσεις, εγώ ταξίδεψα στην Ιορδανία και στο Λίβανο μεταφέροντας και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολιτικές οι οποίες έχουν κάνει κάποιες επιλογές. Παραδείγματος χάρη, επιλογές όσον αφορά, παραδείγματος χάρη, την εξωτερήκευση της ασφάλειας όποιο και να είναι το τίμημα που πληρώνουν οι χώρες αυτές. Και το κόστος για τις χώρες αυτές και για την Τουρκία και για την Ιορδανία και για το Λίβανο είναι ένα πολύ σημαντικό κόστος. Οι χώρες αυτές δεν διάλεξαν τη γεωγραφική τους θέση, δεν έχουν επιλέξει να συνορεύουν με μια χώρα η οποία σήμερα βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση, δεν έχουν επιλέξει να βρίσκονται σε μια Μέση Ανατολή κατεστραμμένη και να πλήττονται από τις συνέπειες μιας πολιτικής χωρίς συνοχή των χωρών μας, καθώς και την δυσκολία να υπάρξει ειρήνη στην κρίση στη Συρία, στον πόλεμο στη Συρία. Θα προσπαθήσω λοιπόν σε τέσσερα σημεία να σας παρουσιάσω τα συμπεράσματά μου. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι παρουσιάσεις που μας έγιναν από τις δύο αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις οποίες ε, εξάλλου ευχαριστώ, με οδηγούν στα εξή συμπεράσματα. Η οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απαραίτητη. Χωρίς αυτή την οικονομική στήριξη δεν μπορούν να καλυφθούν ζωτικές ανάγκες ή ελάχιστες ανάγκες ε, αυτών των ε, ανθρώπων. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να είναι στο ύψος των περιστάσεων, αυτό που θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι είναι απούσα από την πολιτική σκηνή και αυτό είναι κάτι που βεβαίως θα πρέπει να μας απασχολήσει. Η αδυναμία μας, η πολιτική μας αδυναμία και η διπλωματική μας αδυναμία ε, τόπου Όσον αφορά την Ιορδανία, ποιο είναι το δίδαγμα που θα ήθελα εδώ να σας ε, παρουσιάσω. Η έκκληση από μέρους της Ιορδανίας η πολιτική συνεργασία, η πολιτική εταιρική σχέση να είναι στο ύψος της οικονομικής μας στήριξης. Όλοι γνωρίζουν το ρόλο της Ιορδανίας για την ειρήνη στην περιοχή. Διαπιστώνουμε όμως σήμερα ότι οι οικονομικές σχέσεις, οι επενδύσεις, η εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων επενδυτών δεν είναι παρούσα στην περιοχή. Η Ορδανία σήμερα χρειάζεται αυτή τη στήριξη, χρειάζεται τεχνογνωσία και επενδύσεις. Είναι η προϋπόθεση για να υπάρξει συνοχή στην χώρα αυτή. Να υπάρξει κοινωνική συνοχή στην Ιορδανία. Για το Λίβανο θα ήθελα να πω ότι γύρισα με μεγάλες ανησυχίες. 6 εκατομμύρια κατοίκους έχει ο Λίβανος, 2 εκατομμύρια πρόσφυγες συμπεριλαμβανομένων και των ε, Παλαιστίνιων προσφύγων στην Ευρώπη, φοβόμαστε την αποσταθεροποίηση μιας μαζικής ε, εισρωής προσφύγων. Φανταστείτε τι σημαίνει λοιπόν δύο εκατομμύρια πρόσφυγες για μια κοινωνία η οποία πέρασε από 9% ανάπτυξη σε αρνητική ανάπτυξη σήμερα με το 20% του πληθυσμού να ζει κάτω από το επίπεδο φτώχειας με έναν εμφύλιο πόλεμο ο οποίος βρίσκεται πολύ κοντά και με μια συνοχή, κοινωνική συνοχή η οποία πραγματικά είναι εξαιρετικά ασταθής. Εάν ο Λίβανος δεν επανέλθει στην οικονομική ανάπτυξη, πολύ φοβάμαι ότι θα ξεκινήσει μια πάρα πολύ επικίνδυνη εποχή. Οι κρατικές δομές ε, της χώρας αυτής είναι εξαιρετικά αδύναμες και όλος ο δημόσιος τομέας ασταθής. Και βεβαίως ε, με όλο το σεβασμό προς την Αφρική όταν κοιτάω το τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή ε, και στο Λίβανο συγκεκριμένα, πολύ φοβάμαι ότι οδηγούμαστε προς μια κατάσταση που πολύ μοιάζει με την κατάσταση που επικρατεί στην Αφρική. Είναι δηλαδή εξαιρετικά ανησυχητική η κατάσταση στο Λίβανο και θα πρέπει σίγουρα και εμείς να αναλάβουμε τις ευθύνες μας από δημοσιονομικής πλευράς. Η κυρία Κανεμάκη matkalta ja erityisesti mieleen on tietysti... Ευχαριστώ. Από αυτό το ταξίδι γνωρίζαμε πολλά πριν πάμε, αλλά όταν βλέπει κανείς με τα ίδια του τα μάτια τον εντυπωσιάζει η καθημερινή ζωή των προσφύγων. Ήταν αδέκαστος ο ήλιος και η ζέστη, έλειπαν το νερό, τα τρόφιμα, τα ρούχα, έλειπαν τα πάντα. Επιπρόσθετα, θα ήθελα να κάνω μια σύγκριση γιατί εγώ μπόρεσα να πάω και στην Τουρκία με την προηγούμενη υποστολή και εκεί επισκεφθήκαμε κάποιους καταβλισμούς προσφύγων και εκεί η κατάσταση ήταν φρικτή. Όμως αν συγκρίνουμε βάσει τις εμπειρίες που είχαμε εμείς ε, σε αυτά τα δύο ταξίδια μιλάω δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω όλα κριτήρια, αλλά βάσει της εμπειρίες που έχω από αυτές τις δύο επισκέψεις. Μπορώ να πω ότι οι καταβλισμοί στο Λίβανο και στην Ιορδανία ήταν σε πολύ χειρότερη κατάσταση από ότι αυτή στην Τουρκία. Και επίσης, μας ε, το είχαν πει και οι εξωματούχοι των Ηνωμένων Εθνών ότι υπήρχαν προβλήματα βίας, παραδείγματος χάρη, και κάποιες άλλες καταστάσεις που δεν τις συναντάμε τόσο στους καταβλισμούς στην Τουρκία. Όμως εμείς ε, στην Ευρώπη έχουμε ασκήσει μεγάλη κριτική στην Τουρκία γιατί ακόμα τα χειρίζεται τους πρόσφυγες ε, και δεν έχουμε επικρίνει τόσο αυτές τις άλλες χώρες. Πρέπει να πω ότι η βάση της εμπειρίας μου και του ταξιδιού μου ίσως υπερβάλαμε στην κριτική που ασκήσαμε στην Τουρκία γιατί η κατάσταση είναι χειρότερη αλλού. Ναι, πρέπει να επικρίνουμε την Τουρκία, αλλά δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι στο Λίβανο και στην Ιορδανία είναι πολύ χειρότερη η κατάσταση. Όπως και να έχει, είναι αλήθεια ότι ο Λίβανος ε, έχει υποδεκτεί πολύ περισσότερους πρόσφυγες από ότι όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως ακριβώς γι' αυτό θέλουμε και πρέπει να βοηθήσουμε. Στην πολιτική γειτονία θα πρέπει να έχουμε υπόψη αυτό το θέμα. Επίσης, εμείς φαινόμαστε έτοιμοι να επικρίνουμε τους πάντες και λέμε ότι είναι άσχημα τα πράγματα στις γειτονικέ χώρες. Θα πρέπει να είμαστε βέβαια ικανοί να τονίζουμε, να βλέπουμε την πρόοδο που έχει γίνει στις γειτονικέ χώρες. Όταν ε, έχω κατά νου το Λίβανο, την Ιορδανία, την Τουρκία, είναι χώρες με τρομερά προβλήματα και ακόμη και έτσι πρέπει να αναγνωρίζουμε ότι αυτές οι χώρες υποδέχονται τους πρόσφυγες. Αυτές οι κοινωνίες κάνουν τρομερή προσπάθεια, πολύ μεγαλύτερη από την πλούσια Ευρώπη όπου εμείς ε, τονίζουμε πάρα πολύ ότι είμαστε κοινότητα αξιών. Θα πρέπει να σκεφτούμε λίγο περισσότερο για το πώς μεταφράζονται αυτές οι αξίες στην πραγματικότητα, στην πράξη. Αν σκεφτούμε το μέλλον και τη βοήθεια που χορηγεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, εγώ νομίζω ότι θα πρέπει αυτή η βοήθεια να χορηγείται μέσω από ευρωπαϊκούς θεσμούς και οργανισμούς. Όμως, εμείς δεν έχουμε την εμπειρία, ενώ τα Ηνωμένα Έθνη έχουν και την εμπειρία και το προσωπικό. Αν ε, τους δώσουμε δημοσιονομική βοήθεια, σίγουρα αυτοί θα είναι ικανοί να χειριστούν τα πράγματα. Στους τομείς όπου έχει η εμπειρία Ευρωπαϊκή Ένωση, πολύ καλά, αλλά αν η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε σημείο που πρέπει να δημιουργήσει τους δικούς τη οργανισμούς, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν αυτή είναι η καλύτερη λύση. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να μαθαίνουμε από τα λάθη μας, επομένως πρέπει να βοηθήσουμε μέσω της UNICEF και μέσω των Ηνωμένων Εθνών που κάνουν εξαιρετική δουλειά σε πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις. Εγώ δεν ξέρω αν θα ήταν ε, καλύτερο γιατί αυτό που κάνει ουσιαστικά είναι η ανθρωπιστική δουλειά. Εγώ νομίζω ότι αν το έκανε αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν πολύ δύσκολο. Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η ανάπτυξη που θέλουμε να δημιουργήσουμε στις συνθήκες αυτές, ε, καθώς λείπουν τα πάντα, είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει αυτή η ανάπτυξη. Η έλλειψη εκπαίδευσης με εντυπωσίασε εκεί, έλειπαν τα πάντα, αλλά ταυτόχρονα μας έλεγαν ότι δεν ήξεραν πώς μπορούν να έχουν νέους πόρους και παρά το ότι τους έλειπαν τα πάντα, έπρεπε να αγωνιστούν για να χτίσουν ένα μέλλον. Εγώ νομίζω ότι η Ευρώπη πρέπει να μάθει έτσι ώστε με τους σπόρους που έχουμε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον. Πάντοτε λέμε ότι η βοήθεια δεν πρέπει να είναι μόνο χρηματική, αλλά στην περίπτωση αυτή να λείπουν πολλά χρήματα, χρειάζονται πολλά χρήματα. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Γραμματεία και όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στην αποστολή, όλους τους συμμετέχοντες και τον Πρόεδρο και ευχαριστώ και τους εργαζομένους στην αντιπροσωπεία στο ΑΜΑΝ. Κάνουν καταπληκτική δουλειά. Εγώ μπορώ να πω ότι το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε άλλα μέρη δεν ήταν ίσως τόσο επαγγελματικό όσο σε αυτή την επίσκεψη στο Λίβανο και στην Ιορδανία. Ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να κάνει μια προσπάθεια για να μην επιδεινωθεί η κατάσταση και να μην θέσουμε σε κίνδυνο την ειρήνη. Ο κύριος Φερνάντες λείπει. Έτσι λοιπόν. Ο κύριος ε, Συνοδεινός έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα με προσοχή τα όσα αναφέρατε για την ενημέρωση για το ταξίδι στην Ιορδανία και στο Λίβανο. Ήταν περιστατωμένα και δώσαν μια σαφή εικόνα, όπως και της κυρίας ε, Ευρωβουλευτής, Ευρωβουλευτή προηγουμένως που αναφέρθηκε η δεύτερη που μίλησε μετά από εσά. Ήταν πολύ συγκινητικό αυτό που είπε ότι είδε 17χρονους να κοιτούν στα μάτια και να αναρωτιούνται τι κάνουν εδώ ε, αυτοί. Σαν αντίποδα των όσων αναφέρατε, θα σας πω ότι πριν από ένα μήνα ήμουνα στη Συρία. Επειδή κάνετε περιφερειακά βόλτες στο πρόβλημα, Τουρκία, Λίβανο, Ιορδανία, ναι μεν συμβαίνουν αυτά τα οποία είπατε γιατί πήγα στη, στο Λίβανο, θα σας πω όμως τι συμβαίνει στη Συρία. Όντως, όπως είπε ο προλαλής σας, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ούτε διπλωματία, ούτε πολιτική διότι αν διέθετε διπλωματία και πολιτική θα προσπαθούσε να επιλύσει το πρόβλημα στη βάση του και όχι να επιλύσει τα προβλήματα τα οποία έχει δημιουργήσει η κρίση ή ο πόλεμος. Περιφερειακά, όπως αναφέρατε, Τουρκία, Λιβύη, ε, Λίβανο ή η Ορδανία. τουρκια λιβυη λιβανο η Ιορδανία επισκεφθηκα λοιπον τη Δαμασκό και πολλές πόλεις της Συρίας. Θα ήταν νομίζω πολύ ανθρωπιστικό εκ μέρους της Ένωσης εάν συνέτρεχε στα προβλήματα των νοσοκομείων που πήρα εγώ και είδα παιδάκια 4 και 5 ετών χωρίς πόδια έφηβους 16, 17, 18 χρονών να είναι στο κρεβάτι του πόνου και να μην μπορούν ούτε να κοιτάξουν τη μητέρα του στα μάτια και πολλά άλλα τέτοια περιστατικά και νομίζω ότι ο, ανθρωπισμός τον οποίον επαγγέλεστε θα περίσευε εάν βλέπατε αυτές τις καταστάσεις. Όπως επίσης είδα ανεκτήμητα μνημεία τα οποία είναι στην UNESCO να είναι κατεστραμμένα όπως είναι η Παλμύρα ή όπως είναι η Μαλούλα που επισκέφτηκα. 80% χριστιανοί έχουν φύγει όλοι, έχουν κατεδαφιστεί τα μοναστήρια τους, τα σπίτια τους και προσπαθούν από την τέφρα να αναγεννηθούν. Άρα λοιπόν θα πρέπει το πρόβλημα να μην το βλέπετε μονόπλευρα περιφερειακά, αλλά να το βλέπετε στην ουσία, μέσα στο κέντρο, εκεί όπου αυτή τη στιγμή υπάρχει ο πόλεμος και υπάρχει η κρίση. Ευχαριστώ πολύ. Merci. Σας ευχαριστώ. Συναντήσαμε εκπροσώπους της Ευρώπης στη Συρία και στο Λίβανο. Οι περισσότερες πρεσβείες έκλεισαν από την αρχή της σύγκρουσης. Μόνο η Τσεχία άφησε ανοιχτή την πρεσβεία της. Και σίγουρα η κατάσταση από ανθρωπιστική απόψεως στη Συρία είναι δραματική. Το Χαλέπι έχει καταστραφεί. Τα σύνορα είναι κλειστά. Οπότε στο εσωτερικό της Συρίας υπάρχουν μετακινήσεις πληθυσμών, άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε απόγνωση και η ανθρωπιστική βοήθεια είναι εξαιρετικά περιορισμένη από το καθεστώς. Και αυτό περιπλέκει πολύ ε, περισσότερο τα πράγματα και έχετε απόλυτο δίκιο όταν αναφέρεστε στην δραματική κατάσταση επιτόπου. Η ανθρωπιστική βοήθεια θα πρέπει να μπορεί να φτάνει στο πληθυσμό, στους πολίτες στη Συρία που έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Ο κύριος Μπέγκε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παρουσίαση στην οποία εντάξατε και πολλές ενδιαφέρουσες ε, προτάσεις που ε, συνάγεται από τα όσα είδατε και εσείς και οι συνάδελφοί μας εκεί και που έχουν βέβαια και άμεση σχέση και με, την, ε, με τα όσα ακούσαμε στην επίσκεψή μας στην Τουρκία και που οι συνάδελφοί μας είπαν επίσης πολλά και σημαντικά πράγματα τα οποία δεν επιθυμώ να επαναλάβω τα ακούσατε και εσείς να μου επιτρέψετε μόνο να θίξω δύο-τρία θέματα που απορρέουν κιόλας από το γεγονός ότι έχουμε και μπροστά μας οι διαδικασίες σχετικές με τον προϋπολογισμό. Πράγματι, οι χώρες αυτές που βρίσκονται στην άμεση γειτονία της Συρίας, οι χώρες αυτές λοιπόν αντιμετωπίζουν μια τεράστια πρόκληση και στο τέλος της γραφής οφείλουμε να αναγνωρίσουμε, το είπαν και κάποιοι συνάδελφοί μας, ότι οι χώρες αυτές πράττουν περισσότερα από όσα είναι διατεθειμένες να πράξουν οι ίδιες οι χώρες μέλη τη Ένωση. Ας σταθούμε λοιπόν μια στιγμή να σκεφτούμε πού έχουν πάει αυτές οι κοινέ αξίες που υποτίθεται ότι αποτελούν τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν εξετάσουμε πώς διαμορφώνεται η χρηματοδότηση των διαφόρων αυτών μέτρων. Έχω να πω το εξής. Άκουσα ότι μέχρι το φθινόπωρο, λόγω των διάφορων δραστηριοτήτων όπου έχουμε και εμείς συμμετάσχει στις διάφορες διαδικασίες, μέχρι το φθινόπωρο λοιπόν, με τις υποσχέσεις που έχουμε δώσει εφόσον αυτές υλοποιηθούν, τα βγάζουμε πέρα. Όμως έχουμε και τις εμπειρίες από το 2014 και μετά. Και αυτό μας οδηγεί να σκεφτούμε ότι πρέπει ήδη να φροντίσουμε και για τις ανάγκες του 2017. Να μην φτάσουν τα παιδιά το φθινόπωρο να μην μπορούν να πάνε στο σχολείο διότι δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα. Γίνεται στην Τουρκία τώρα συνάντηση των ε, χωρών που συμμετέχουν στις χρηματοδοτήσεις αυτές και που εκεί συζητούνται και οι χρηματοδοτικές ανάγκες. Να σας δώσω νούμερα το Ταμείο Κατεπικουσών Αναγκών των Ηνωμένων Εθνών είναι κατά 70% εκατομμύρια, συγγνώμη, 70 εκατομμύρια χαμηλότερο από αυτό που προβλεπόταν τον προηγούμενο χρόνο. Πρέπει να φτάσουμε να ευθυγραμμίζονται οι υποσχέσεις με το σχεδιασμό. Οι υποσχέσεις δηλαδή για χρηματοδοτήσεις. Άλλωστε είναι σημαντική η συμμετοχή του κοινοτικού προϋπολογισμού στη χρηματοδότηση που προσφέρουν τα Ηνωμένα Έθνη. Αυτά τα θέματα πρέπει να συζητηθούν στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Και κυρίως πρέπει να επιβεβαιωθούν οι υποσχέσεις που έχουν δοθεί. Δηλαδή, να μην ερχόμαστε ξανά σε νέες διαδικασίες κατεπίγοντος χαρακτήρα που οδηγούν σε κατασπατάληση του χρόνου για να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες που είναι προφανές ότι πρόκειται να προκύψουν. Και έχουμε και τη γνωμοδότηση για την αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου για τα διάφορα ταμεία, ταμεία κατεπηγουσών αναγκών, για το Ταμείο Αφρικής κλπ. Που βρίσκονται σε πολύ περιορισμένο επίπεδο. Και οι συνεισφορές παραμένουν στα ελάχιστα επίπεδα. Με την ελπίδα ότι οι εθνικές ανθρωπιστικές οργανώσεις θα λάβουν το μεγαλύτερο δυνατό μέρος της πίτας. Από αυτή την περιορισμένη χρηματοδότηση. Δεν είναι δυνατόν. Αν δεν αλλάξουν τα πράγματα αυτά, εγώ πάντως δεν πρόκειται να συμφωνήσω ξανά με τέτοια outsourcing ταμείων. Δεύτερο ερώτημα που προκύπτει στα μάτια μου, σε ό,τι αφορά την, τον μέσο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, εκεί πρέπει να κάνουμε κάθε τι το δυνατόν για να επιτύχουμε ώστε χώρες που αντιμετωπίζουν τέτοια πίεση, όπως οι χώρες αυτές που επισκεφθήκατε, Ιορδανία, Λίβανος, και ανεξαρτήτως των εσωτερικών προβλημάτων που συνεπάγονται όλα αυτά, χώρες που βρίσκονται στη γειτονία μας, και ορισμένε από αυτέ είναι και αποτυχημένε χώρε είναι failed states. Πού, πώς θα μπορέσουμε να τις ενισχύσουμε. Αυτό έχει σχέση και με την ετήσια χρηματοδότηση και με την αναθεώρηση του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου, αλλά και με το ερώτημα ποια θα είναι η στρατηγική προσέγγιση για την χρηματοδότηση αυτή. Διότι μέχρι τώρα δεν έχουν εξασφαλίσει οποιαδήποτε σταθεροποίηση τα χρήματα που έχουμε διαθέσει στις χώρες αυτές. Και τώρα ζούμε το εξή. Έχουμε τη διαδικασία για τον προπολογισμό του 2017, αναλύσεις για το προσφυγικό, που είναι πραγματικά εξαιρετικά περίπλοκες και οδήγησαν τελικά σε καθυστέρηση υποβολής του προσχεδίου προπολογισμού πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βλέπουμε από την άλλη μεριά ανακοίνωση τη κυρία Μογκερίνη, που μαζί με τον Φραν αρχές Ιουνίου από ό,τι φαίνεται προτίθεται να κάνει μια ευρία πρόταση η οποία θα αναφέρεται ιδίω σε ανάγκες σημαντικών επενδύσεων στην Βόρεια Αφρική αλλά και σε άλλες γειτονικέ χώρες της Ευρώπης και πέραν αυτού θα αναφέρει και σχετικά με χρηματοδοτικές συμβολές μετακίνηση πιστώσεων για να αντιμετωπιστούν θέματα μετανάστευσης και προσφυγικού. Πράγματα τα οποία είχαν ήδη συζητήσει και είχαν θέσει στην πολιτική συζήτηση συναδελφοί μας και τα τελευταία. Εντυπωσιάζομαι λοιπόν από την ευελιξία που δείχνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά από αυτήν προκύπτει τώρα η εξή ερώτηση. Όταν έρχεται η κυρία Μογκερίνη και ανακοινώνει αρχές Ιουνίου, δηλαδή θα περιμένει το βρετανικό δημοψήφισμα και καλά θα κάνει. Θα κάνει λοιπόν τις προτάσεις αυτές, λέει, τότε εγώ λέω ότι ελπίζω ότι και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη συνάντηση κορυφής του 28 Ιουνίου θα αποδεχτεί τις προτάσεις της αυτές. Και ξαναμπαίνουμε στο παλιό παιχνίδι. Τα είπα πριν αυτά και στην Επιτροπή Ίντα. Το Συμβούλιο αποφασίζει. Αν δεν αποφασίσει, τότε ίσως πρέπει το Κοινοβούλιο να στραφεί κατά του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. διότι αλλιώς μπορούμε να το κλείσουμε το μαγαζί και να πάμε σπίτια μα. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι θέλουμε να επιτρέψουμε κάτι τέτοιο ή μέσα στις χρονικές διαδικασίες μέχρι τις 28, 28 συγγνώμη, έκτου υπάρχει δυνατότητα να γίνουν και κάποιες προκαταρκτικές συζητήσεις με το Συμβούλιο ώστε να ακολουθεί και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, να παρακολουθεί τη διαδικασία αυτή και το Κοινοβούλιο ή και να χρησιμοποιήσουμε τις συναντήσεις που έχουμε μέχρι τότε ώστε να λάβουμε θέση, να τοποθετηθούμε απέναντι στις εξελίξεις αυτές. Διότι ενδεχομένως να υπάρξει απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου όπου εμείς θα είμαστε απλώς κομπάρσι. Θέλω λοιπόν να θέσω το θέμα, να συζητήσουμε τα όσα προτίθεται να βράξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε, όπως είπα, να είναι ενεργός ο ρόλος και συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ. Merci. Ευχαριστώ. Σήμερα το απόγευμα θα επανέλθουμε στο θέμα των τροπολογιών των συναδέλφων. Και αν καταλαβαίνω καλά, η ψηφοφορία θα γίνει τέλος Ιουνίου, μάλλον. Η κυρία Μυριάντα. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που ήταν σε αυτή την αποστολή γιατί νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερο να αντιληφθεί κανείς τι γίνεται επί τόπου εάν μπορέσει να επισκεφθεί και να δει πραγματικά όλα αυτά που κάνουμε εδώ πώς ε, επηρεάζουν, τι συνέπειες έχουν για τους ανθρώπους αυτούς επιτόπου. Το θέμα της εκπαίδευσης, πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι χτίζονται οι απαραίτητες δομές, βιώσιμες δομές για να προσφέρουν ε, εκπαίδευση, παιδεία σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, καθώς και σε κάποιες ε, άλλες δομές που χρειάζονται οι συζητήσεις συνεχίζονται. Και πραγματικά δεν βλέπω βιώσιμες λύσεις. Θα πρέπει να έχουμε μία λίγο πιο μακροπρόθεσμη ε, πολιτική και να δούμε πώς αυτά που αποφασίζονται εδώ υλοποιούνται επί τόπου. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Σας ευχαριστώ, κυρία Μυριάντα. Ξέχασα να αναφερθώ και στον Σίκφριντ Μούρεγαν που ήταν επίσης παρόν στο ταξίδι. Σας ευχαριστώ για αυτά που είπατε. Όλοι όσοι πήρατε το λόγο, είτε ήσασταν μαζί μας είτε όχι. Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε εδώ το πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση και βεβαίως θα προετοιμάσουμε και μία αναφορά, μία έκθεση η οποία θα υποβληθεί σε κάποια μελλοντική μας συνάντηση. Εγώ ήδη έχω προετοιμάσει κάποια από αυτά που θέλω να μπουν στην έκθεση και τα έχω βάλει στον ιστότοπο της Επιτροπής και πολλοί άλλοι όμως ακούγοντάς σας διαπιστώνω ότι θα πρέπει να προσθέσετε σε αυτήν την παρουσίαση που θα κάνουμε της ε, αποστολής μας, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε μία κίνηση. Δεν μπορεί κανείς να πει και συμφωνώ εδώ με τον κύριο Μπέγκε ότι στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο μειώσαμε τα κονδύλια που απευθυνόταν ε, σε αυτήν την πολιτική και την πολιτική των μεταναστών και των προσφύγων ενώ το 2011, το 2012 υπήρχαν παρόμοια φαινόμενα. Δεν ήμασταν λοιπόν αρκετά προνοητικοί. Η κρίση αυτή δεν πρόκειται να σταματήσει τα επόμενα χρόνια και οι συνέπειες για την Ευρώπη είναι πάρα πολύ σημαντικές. Εάν η Ευρώπη λοιπόν θέλει να παραμείνει πιστή στις αξίες της, αυτές οι καταστάσεις είναι εξαιρετικά σοβαρές για τις ευρωπαϊκές αξίες. Και μάλιστα πήγαμε να επαληθεύσουμε και να ελέγξουμε κι εμείς αυτά που στις 10 Μαΐου μας ανακοίνωσε η κυρία Μογκερίνη, η οποία ανακοίνωσε ότι μόλις ε, ληφθούν κάποιες αποφάσεις όσον αφορά χρηματοδότηση, αυτό μεταφέρεται επιτόπου σε δράση βλέπουμε ότι το 80% των ε, κονδυλίων που μεταφέρονται στα κράτη-μέλη πίσω σαν τα μία ε, κονδύλια συνοχής ουσιαστικά μας αφήνουν εντελώς ακάλυπτους όταν προκύψει μια τέτοια κρίση και η Ευρώπη δείχνει σε μια τέτοια περίπτωση πόσο ανίσχυρη είναι. Όλοι οι πρόσφυγες, τους οποίους συναντήσαμε, μας είπαν ότι θέλουν να γυρίσουν στις χώρες τους και αυτό δεν μπορεί να γίνει αν δεν υπάρξει ειρήνη στη Συρία. Ήμασταν τη Δευτέρα το βράδυ χωρισμένοι σε δύο διαφορετικές ομάδες και στην επιστροφή μας προς το Αμάν σταματήσαμε σε ένα προάστιο το Ζάρκα. Η μία από τις δύο ομάδες πήγε σε ένα κτίριο και ανεβήκαμε 82 σκαλιά, 5 πέμπτο όραφο. Ήταν μια οικογένεια από τη Συρία με έξι παιδιά με ειδικέ ανάγκες. Πρόκειται για ένα κτίριο χωρίς ασανσέρ. Ανεβαίνουν δηλαδή καθημερινά πέντε ορόφους με τα πόδια. Ο πατέρας αυτής της οικογένειας μας ρώτησε τι κάνει η Ευρώπη ακριβώς για να σταματήσει αυτή η σφαγή παιδιών αλλά και ενηλίκων στη Συρία. Σήμερα όλοι συμφωνούμε ότι δεν μπορεί παρά να υπάρξει πολιτική λύση. Και το ερώτημα είναι αν η Ευρώπη συμμετέχει στην εξέβρεση αυτής της πολιτικής λύσης. Γιατί βλέπουμε το ρόλο που παίζει ο Πούτιν, το Ιράν, οι Ηνωμένε Πολιτείε, οι χώρε του κόλπου που χρηματοδοτούν τον εξοπλισμό, τους εξοπλισμούς επιτόπου. Τι κάνει όμως ακριβώς η Ευρώπη. Αυτό είναι το ερώτημα. Πέραν δηλαδή της ανθρωπιστικής βοήθειας, βρισκόμαστε στην αρχή του 21ου αιώνα και ίσως η Ευρώπη θα πρέπει να εκφράσει μεγαλύτερη πολιτική φιλοδοξία. Και ισχύει. Και αυτό βεβαίως είναι κάτι που σίγουρα θα πρέπει να συζητηθεί εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ελπίζω όλοι να μπορέσουμε να παίξουμε ένα ρόλο, να μην περιμένουμε δηλαδή το Συμβούλιο και να παραμείνουμε απλώς ο αρμόδιος για την καταγραφή των αποφάσεων του Συμβουλίου. Αυτά όσον αφορά το θέμα. Αυτό ήταν ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Σας ευχαριστώ όλους για την παθιασμένη σας συμμετοχή. Ευχαριστώ και τη Γραμματεία της Επιτροπής για την στήριξή της μέχρι τώρα και για την προετοιμασία που θα κάνει για την έκθεση που θα υποβάλουμε. Και τώρα θα προχωρήσουμε στον διορθωτικό προϋπολογισμό για το 2016. Το δεύτερο σχέδιο προϋπολογισμού είναι αυτό. Ο Χωσέ Μανουέλ Φερνάντες δεν είναι σήμερα εδώ και μου ζήτησε Μου ζήτησε να αναλάβω εγώ αυτή την αποστολή που μου αγγίζει πάρα πολύ, αλλά και μπορώ να πω ότι μου προκαλεί και άγχος, γιατί θα αντικαταστήσω τον ε, γενικό εισηγητή μας για τον ε, προπολογισμό του 2016. Πρόκειται για ένα σχέδιο ορθικού προπολογισμού την Άνοιξη. Εδώ θα πρέπει να περιμένουμε γιατί η Κομισιόν ε, θέλησε ουσιαστικά να διορθώσει αυτές τις προβλέψεις ε, για την υποδοχή των προσφύγων και μεταναστών και δεν θα μπορέσει να μας κάνει προτάσεις ε, αυτές οι Κομισιόν παρά στα τέλη Ιουνίου. Έτσι λοιπόν ε, έχουμε τώρα προβλέψεις του καλοκαιριού και όχι της άνοιξης. Αυτό που μας προτείνει η Κομισιόν βάσει προσωρινών οργανισμών του 2015 που καταρτίστηκαν στις 31 Μαρτίου του 2006 να, βάλουμε στον προπολογισμό του 2006 το πλεόνασμα από το οικονομικό ε, του 2015 του 1,3 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό σημαίνει μείωση των εθνικών συνεισφορών στον προϋπολογισμό. Πρόκειται για κάτι ιδιαίτερα ευχάριστο λοιπόν για τους εθνικούς προϋπολογισμούς, αλλά δεν έχει κανένα αντίκτυπο στο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως σε αυτό το στάδιο ίσως θα ήταν καλό να δώσω το λόγο στον κύριο Σιλβάνο Πρέσα, ο οποίος είναι γενικός διευθυντής της δεύτερης της ε, Κομισιόν, για να μας παρουσιάσει σε γενικές γραμμές αυτό το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού υπαριθμών 2 και κατόπιν ε, θα σας πω τι μας προτείνει να υιοθετήσουμε ο κύριος ε, Φερνάντες. Παρακαλώ κύριε Πρέσα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όσο αναφέρατε, πρόκειται εδώ για με ένα κλασικό διορθωτικό προϋπολογισμό που προβλέπεται στο άρθρο 18 του χρηματοοικονομικού κανονισμού και θα πρέπει να παρακτεί τουλάχιστον 15 μέρες, το αργότερο 15 μέρες μετά την υιοθέτηση των προσωρινών λογαριασμών που παρουσιάστηκαν στα τέλη Μαρτίου. Το πλεόνασμα που παρουσιάζεται και θα πρέπει να εγγραφεί στον προπολογισμό ακολουθεί μια μεθοδολογία που υπάρχει στον κανονισμό για τους ίδιους πόρους. Το επεξηματικό μήνυμα που ε, συνοδεύει το σχέδιο του προπολογισμού, μας ε, δίνει πώς γίνεται ο υπολογισμός και την προέλευση του πλεονάσματος. Έτσι λοιπόν, στον πρώτο πίνακα που περιλαμβάνεται στην ε, αιτιολόγηση του σχεδίου προπολογισμού, το σημείο αφετηρίας ε, είναι η διαφορά στην ισορροπία μεταξύ των δαπανών και των εισόδων. Αν δούμε τις ε, πληρωμές που έγιναν το 2015, τις εκταμιεύσεις που έγιναν και το συγκρίνουμε με το εισόδημα που ελήφθη κατά τη διάρκεια του έτους, κατόπιν λαμβάνει υπόψη την ακύρωση των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το 2014 στο 2015 και αυτή η ακύρωση λαμβάνεται υπόψη αν δεν έχει χρησιμοποιηθεί πλήρως και επίσης λαμβάνει υπόψη τις πιστώσεις υποχρεώσεων που είχαν εγγραφεί στον προπολογισμό του 2015 και μεταφέρθηκαν στο 2016. Γιατί αυτά τα χρήματα παραμένουν στα βιβλία και μας επιτρέπουν την ολοκλήρωση της εφαρμογής σύμφωνα με τις συνθήκες που προβλέπονται στο χρηματοοικονομικό κανονισμό. Το αποτέλεσμα αυτής της μεθόδου υπολογισμού είναι πράγματι ένα πλεόνασμα 1,3 δισεκατομμυρίων. Τα τρία τέταρτα σχεδόν προέρχονται από τα έσοδα και το 1 τρίτο προέρχεται, το ίμιση αυτού του 1 τρίτου προέρχεται από πρόστιμα που έγιναν οριστικά μετά τον ε, τελευταίο διορθωτικό προπολογισμό του 2015 και ένα άλλο τμήμα είναι η μη εφαρμογή των δαπανών, η στην απορρόφηση. Και εδώ βλέπετε το δεύτερο πίνακα που εξηγείται στο σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού. Το περισσότερο, το μεγαλύτερο μέρος του πλεονάσματος σχετίζεται με τους ίδιους πόρους και αυτό έχει να κάνει με παραδοσιακούς πόρους, το ΦΠΑ και από το καθάριση των χωρίς εισόδημα και εδώ έχουμε και ένα στοιχείο που πλήττει το αποτέλεσμα και είναι η συναλλαγματική τιμή όταν συνελέχθηκαν, τιμή του όταν συλλέχθηκαν οι πόροι. Τακτικά συλλέγονται και οι εισφορές το καθαριστό χωρίς οδήματος στέλνονται μηνιαία και καταβάλλονται σε εθνικά νομίσματα. Έτσι λοιπόν τα κράτη-μέλη που είναι εκτός Ευρωζώνης ε, πληρώνουν στο εθνικό τους νόμισμα και κατόπιν μεταφράζεται σε ευρώ ανάλογα με τη συναλλαγματική ισοτιμία του μήνα. Έτσι λοιπόν αυτό προκάλεσε κάποιες διαφοροποίησεις με τις αρχικές εκτιμήσεις και αυτό προκαλεί μια διαφορά μεταξύ των αρχικών εκτιμήσεων και του αποτελέσματος του τέλη του έτους. Εδώ επίσης παρεμβαίνει ο περιπολογισμός που γίνεται τη ίος, της έκπτωσης του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό γίνεται σε μία πενταετή περίοδο και έτσι λοιπόν ε, και εδώ η συναλλαγματική ισοτιμία μπορεί να έχει αντικτύπω στο αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν όλα αυτά μας οδηγούν στα τρία τέταρτα του πλεονάσματος που προέρχεται από τα έσοδα. 180 εκατομμύρια περίπου προέρχονται από τα πρόστιμα και σε ό,τι αφορά τις δαπάνες υπάρχει έχουμε 185 εκατομμύρια που δεν δαπανήθηκαν και τα περισσότερα από αυτά σχετίζονται με τις διοικητικές δαπάνες θεσμικών οργάνων ε, άλλων πέραν της Κομισιόν. Έτσι λοιπόν ε, η Κομισιόν δεν σε 92 εκατομμύρια σε σύγκριση με τα 94 εκατομμύρια για τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα. Ο προπολογισμό της Κομισιόν προς εφαρμογή είναι περίπου 37 φορές μεγαλύτερο από τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα. Έτσι λοιπόν και αυτό εν συντομία εξηγεί τι έχουμε στο σχέδιο ερωτικού προπολογισμού υπαριθμών 2. Εδώ προβλέπεται από το χρηματικό κανονισμό ότι αυτό ο ερωτικό προπολογισμό μπορεί να ασχολείται μόνο με το πλεόνασμα και τίποτα άλλο. Στην ε, γνωμοδότηση θα ήθελα να καλωσορίσω τη σύσταση που γίνεται από τον εισηγητή και η Κομισιόν ελπίζει ότι κατόπιν συμφωνίας στο αρμόδιο φόρουμ στο Συμβούλιο. Ο διορθωτικός προϋπολογισμός μπορεί να προχωρήσει και να, εγκληθεί, να εγκριθεί το συντομότερο. Και αυτό θα δημιουργήσει την ίδια δυναμική που είδαμε και πέρσι στο διορθωτικό προϋπολογισμό. και ίσω ε, να είναι και καλό ιονό για την υπόλοιπη διαδικασία για το σχέδιο προπολογισμού για το 2017. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Διευθυντά. Ευχαριστώ για την ανάπτυξη του θέματο. Μειώσατε το suspense διότι αποκαλύψατε την θέση του εισηγητού την οποία προτιθέμεν, προτιθέμεν θέμη να αποκαλύψω εγώ. Ο κύριος ε, Κονζάλης λοιπόν προτείνει έγκριση του διορθωτικού προϋπολογισμού για το 2016 και απευθύνει έκκληση στις χώρες μέλη να προχωρήσουν σε αυτή την διάθεση του 1,3 δις ευρώ για να σεβαστούν τις ε, υποχρώσεις τους τις ε, υποχρώσεις για το Ταμείο Αφρικής για ε, τα χρήματα που θα δοθούν στην ε, Τουρκία για την αντιμετώπιση του προσφυγικού που ε, εξηγήσαμε διαμακρόν πριν από λίγη ώρα μετά από την επίσκεψή μας στον Λίβανο. Ο κύριος Φερνάντες επιμένει στην ανάγκη να μετρηθεί αυτό στη βάση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος και πέραν του κάθε πλεονάσματος από ενδεχόμενη ε, υστέρηση των ε, εκτελουμένων, κάτω δηλαδή από το περιθώριο που προβλεπόταν. Διότι εν τέλει αυτό που γίνεται είναι να ε, δίνεται το μέρισμα στις χώρες μέλη. Ενώ, ας πούμε, η Γενική Συνέλευση δεν έχει καν ακόμη εγκρίνει τον ισολογισμό. Δηλαδή εδώ βασιζόμαστε σε ένα προσωρινό έγγραφο, στη βάση δηλαδή ενός προσωρινού εγγράφου προχωρούμε χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι στοιχειώδεις αρχές της λογιστικής. Κάπως λοιπόν υπερβολικά γρήγορα διατίθεται τα πλεονάσματα ενώ όπως είπα οι λογαριασμοί δεν είναι ακόμα οι οριστικοί και δεν έχουν ελεγχθεί από το ελεγκτικό συνέδριο σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία τους. Λέγοντας ε, τα λόγια αυτά, ελπίζω ότι απηχώ ε, με ακρίβεια τις απόψεις του εισηγητού. Ποιος επιθυμεί τώρα να λάβει το λόγο. Ουδής. Καλά λοιπόν. Αρκούμεθα σε αυτά τότε. Ε, προφανώς τα όσα εξήγησε ο κύριος Πρέζα ήταν αρκετά πιστικά. Τώρα έχουμε ένα θετικό υπόλοιπο της τάξης των 182 εκατομμυρίων. Ποιες, ε, ε, ε, τι οδήγησε σε αυτά τα πλεονάσματα των ανταλλαγών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτό συνδέεται με την ισοτιμία που εφαρμόζεται στις εθνικές εισφορές όταν αυτές εισπράττονται αναμίνα. Εθνικές εισφορές δηλαδή στη βάση του ΑΕΠ και βασίζονται αυτές σε μια ισοτιμία στην αρχή του, που γίνεται στην αρχή του προϋπολογισμού και μετά για τις χώρες εκτός ζώνης ευρώ καταβάλλονται σε εθνικό νόμισμα και εφόσον η μετατροπή σε ευρώ γίνεται στη βάση της ισοτιμίας της τωρινής μπορεί να κινηθούν προς ε, θετικό πρόσημο ή προς αρνητικό πρόσημο. Εξαρτάται από την ισοτιμία μεταξύ του εθνικού νομίσματος και του ευρώ. Για το 2015 το αποτέλεσμα ήταν ότι η μετατροπή των εθνικών εισφορών, των μηνιαίων ε, εθνικών εισφορών σε ευρώ, απέδωσε ένα θετικό υπόλοιπο. Και όμως ε, ε, ε, ανατιμήθηκε το ευρώ το 2015. εξαρτάται απέναντι σε ποιο νόμισμα εννοείται. Απέναντι στο δολάριο λέει ο πρόεδρος. Χωρίς μικρόφωνο όμως. Και απέναντι στη Στερλίνα, κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά νομίσματα που είναι ακόμη εκτός ζώνης ευρώ. Γίνεται λοιπόν ένας υπολογισμός στη βάση της μεθόδου που σας ανέπτυξα και με τον επανυπολογισμό της Βρετανικής Επιστροφής η οποία επανεξετάζεται κάθε χρόνο στη βάση της προηγούμενης τετραετίας. Ο συνδυασμός όλων αυτών αποδίδει αυτό το αποτέλεσμα που όπως είπα ε, εξαρτάται από την ισοτιμία και για την χρήση του 2015 οδήγησε σε ε, θετικό υπόλοιπο 180 ε, εκατομμυρίων. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, όσον αφορά το σχέδιο του διαθετικού κομπλισμού 2, ολοκληρώνεται η συζήτηση. Η τελική έκθεση θα υποβληθεί για ψηφοφορία ή 15 ή 16 Ιουνίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή ή 15 ή 16 Ιουνίου και ενδεχομένως η ψηφοφορία στην Ολομέλεια θα λάβει χώρα στις 6 Ιουλίου. Προθεσμία υποβολής τροπολογιών 26 Μαΐου. Μεθαύριο δηλαδή. Και τώρα θα δώσουμε το λόγο στον συνάδελφο τον κύριο Νεγκρέσκου ο οποίος είναι εισηγητής για την κινητοποίηση του Ταμείου Προσαρμογής για την Παγκοσμιοποίηση. NO Machinery. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόκειται για μια πρόταση τη του Βελγίου, 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα ποσό για την κάλυψη του προβλήματος που έκυψε στη Βαλονία, την εταιρεία ΕΝΟ, για το σχέδιο ΕΝΟ, 88 άτομα τα οποία απολύθηκαν από την κατασκευαστική αυτή η εταιρεία. Πρόκειται για μια εταιρεία στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Πρόκειται για ένα μεγάλο μέρος νέων, νέων οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση σε άλλες ε, θέσεις απασχόλησης και το ποσό αυτό θα πρέπει να στηρίξει τους ανθρώπους αυτούς για να μπορέσουν να εποφεληθούν από επαγγελματική κατάρτιση. 3 εκατομμύρια ευρώ είναι το συνολικό ποσό και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση θα στηρίξει με 1,8 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή λίγο παραπάνω από το 50% του συνολικού ποσού. Υπευλήθη το πρώτο αίτημα στις 7 Δεκεμβρίου του 2015. Αρχικά η εταιρεία ήταν η Caterpillar με διάφορους ε, άλλους ε, εταίρους στην περιοχή η έλλειψη ανταγωνιστικότητας αλλά και η φυγή κάποιων επιχειρήσεων που μετατοπίστηκαν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης οδήγησε στην κατάσταση αυτή. Πρόκειται λοιπόν για την συνέχεια ενός ε, προγράμματος που είχε ξεκινήσει το 2014, μάλλον το 2013 και αφορούσε 1.400 εργαζόμενους που έχασαν τη δουλειά τους. Πρόκειται δηλαδή για μια περιοχή που έχει πληγεί πολλαπλά τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό και θέλουμε το Ταμείο αυτό προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση να στηρίξει αυτό το σχέδιο και βεβαίως περιμένουμε τις προτάσεις σας ε, εφόσον έχετε. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν παρατηρήσεις. Ο κύριος Ντενανό. Έχουμε ελέγξει εάν ε, η στήριξη αυτή είναι συμπληρωματική των εθνικών ε, δυνατοτήτων χρηματοδότησης. Ναι, αυτό το πρόβλημα υπάρχει. Πάντα. Δηλαδή, από ό,τι μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εδώ τηρούνται οι αρχές που διέπουν το Ταμείο αυτό προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση, δηλαδή το 50% χρηματοδοτείται από το Βέλγιο. Δεν έχω βεβαίω συγκεκριμένα στοιχεία και ενδεχομένως η Επιτροπή να μπορεί να μας πει κάτι γι' αυτό. Ευχαριστώ η Επιτροπή. Εγώ πρέπει να σας πω ότι στη δική μου χώρα, από ό,τι ξέρω, πρόκειται για ένα τρόπο να χρηματοδοτήσουν ε, κάπως ε, τα κράτη-μέλη και τους δικούς τους προπολογισμούς. Εσύ κύριε Διευθυντά, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, αυτό εντάσσεται στους όρους επιλεξιμότητας. Ε, να ληφθεί υπόψη δηλαδή, να ληφθούν υπόψη και οι εθνικοί μηχανισμοί και εφόσον η κινητοποίηση αυτή είναι συμπληρωματική των εθνικών μηχανισμών και δεν τους υποκαθιστά και εφόσον αυτοί ε, εξυπηρετούν, ε, ε, στηρίζουν δηλαδή τους εργαζομένους οι οποίοι έχουν απολυθεί. Ευχαριστώ για την απάντησή σας που δεν ε, αποκλείει και άλλες ερωτήσεις. Θα αρκεστούμε σε αυτά. Αν δεν υπάρχουν άλλοι που επιθυμούν να υποβάλουν ερωτήσεις, οι τροπολογίες θα πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι τις 2 Ιουνίου θα επανέλθουμε στις 15 Ιουνίου έκτου δηλαδή για να ψηφίσουμε θα εγκρίνουμε τότε την έκθεση και στις 23 έκτου θα φτάσει το έγγραφο στην Ολομέλεια. Κυρία Μούντι θα ακολουθήσει, που θα έπρεπε κανονικά να της δώσω αμέσω το λόγο. Έχουμε όμως τον κύριο Ροζεύσκη που είναι επικεφαλής αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με το Λευκορωσικό Κοινοβούλιο και που είναι υποχρεωμένος να εγκαταλείψει την αίθουσα στις 12.30 το αργότερο. Δέχεστε, απρόκειται για την ε, κατεξουσιοδότηση πράξη για την ε, Λευκορωσία κλπ. Μήπως μπορούμε κυρία Μούντι να δούμε το θέμα σας μετά. Ναι, αλλά ε, μέσα, μέσα στο σημερινό πρωινό ε, στην σημερινή πρωινή συνεδρίαση, κύριε Πρόεδρε. Ναι, σας ευχαριστώ λοιπόν για την κατανόηση που δείχνετε. Η Επιτροπή Προϋπολογισμών, ως γνωρίζετε, αναμένει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις αποφάσεις της 15ης ε, Τετάρτου, οι οποίες προσθέτουν την ε, Λευκορωσία στις χώρες που μπορούν να επωφεληθούν από εγγυήσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για δάνεια τα οποία χορηγεί στην Λευκορωσία. Έχουν προσκληθεί μετά από ενημέρωσή τους οι βουλευτές της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, δε κύριος Σδρογεύσκη, που είναι επικεφαλής της αντιπροσωπείας για σχέσεις με το Λευκορωσικό Κοινοβούλιο και είναι σήμερα παρόν και τον ευχαριστώ. Επίσης παρόν είναι ο κύριος Μέρεντιθ επικεφαλής της διεύθυνση για Σχέσεις Γειτονίας και Διεύρυνσης και ο Τιματάρχης για τις σχέσεις με την Τράπεζα ε, Επενδύσεων, με την Τράπεζα Νοικοδόμησης και άλλα πρόσωπα που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και στην Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων. Εάν επιθυμείτε λοιπόν, μπορώ, αν συμφωνείτε μάλλον, μπορώ να δώσω το λόγο στην κυρία Γουάρια Ζαμπάλ που είναι η διαρκής εισηγήτριά μας για θέματα ε, τράπεζας επενδύσεων. Ευχαριστώ Πρόεδρο. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε και την ευκαιρία να ακούσουμε τους προσκεκλημένους σε αυτή τη συζήτηση. Όταν η Κομισιόν μας έστειλε αυτή την πρόταση, η ομάδα FTD εξέφρασε κάποιες αμφιβολίες και συζήτησε το θέμα του να θέσουμε μια αντίρρηση σε αυτές τις κατοσυγκροτήσεις και εμείς ε, ως συντονιστές ε, σκεφτήκαμε ότι θέλουμε να λάβουμε όσο δυνατόν περισσότερες πληροφορίες. Γι' αυτό έχουμε αυτούς τους προσκεκλημένους. Βεβαίως, ε, εξαρτάται από ποια σκοπιά βλέπει κανείς το ζήτημα. Σίγουρα μπορεί να υπάρχουν ε, κάποιες αμφιβολίες ε, για την δημοκρατική ποιότητα μιας χώρας για τους ε, θεσμούς της. Όμως, αν απορριφθεί η βοήθεια σε αυτές τις χώρες, ουσιαστικά πλήττει αρνητικά και τους πολίτες. Και το ίδιο συμβαίνει και με σχέδια συνεργασίας. Τελικά οι πολίτες είναι αυτοί που θίγονται περισσότερα και φυσικά αυτούς παντού προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Να δούμε λοιπόν ποιες θα είναι οι πληροφορίες που θα μας δώσουν τα μέλη της Επιτροπής σε αυτή την περίπτωση και ο πρόεδρος της Αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Ένωσης Λευκορωσίας. Για θα προσπαθήσουμε να λάβουμε την καλύτερη δυνατή απόφαση σε αυτή την Επιτροπή. Ευχαριστώ. Θα ζητήσω από τον Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας να πάρει το λόγο, κ. Σοζεύσκη. Παρακαλώ, μπορείτε να μας πείτε την άποψή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Ευχαριστώ που ζητήσατε να ακούσετε τη γνώμη μας. Δεν θα με Αναφέρομαι βασικά σε τρία στοιχεία. Πρώτο, το αντικείμενο, δηλαδή η κατεξουσιοδότηση στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Απριλίου, γενικά είναι ορθά συνταγμένη. Προβαίνει σε μια σωστή διάγνωση της καταστάσεως στην Λευκορωσία. Τονίζει επίσης ότι οφείλει να ληφθεί η απόφαση περί της οποίας πρόκειται. Περιγράφει δε την κατάσταση με τέτοιο τρόπο ώστε να προκύπτει ότι είναι σωστό να ληφθεί απόφαση. Το ε, έγγραφο είναι σωστά συνταγμένο και περιλαμβάνει τα στοιχεία εκείνα που είναι απαραίτητα για την λήψη αποφάσεως. Δεύτερο, εγώ τάσομαι υπέρ τη ε, συνεργασία με την Λευκορωσία και μάλιστα πρέπει να ενισχυθεί η χώρα αυτή και σε ό,τι αφορά τις υποδομές. Σε κάθε δε φάση της συνεργασίας πρέπει να μετρείται η πρόοδος. Υπενθυμίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάθε επανάληψη έχει τονίσει ότι η κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην ε, Λευκορωσία πρέπει οπωσδήποτε να βελτιωθεί. Η διαδικασία για την καταχώρηση των υποψηφίων των κομμάτων πρέπει επίσης να βελτιωθεί μέσα σε αυτήν την ε, προσπάθεια. Και βεβαίως η λειτουργία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Οι, ε, οι τελευταίοι μήνες στη Λευκορωσία αποδείχνουν ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα από την απόψη αυτή. Επιβάλλονται χρηματικές ποινές και πρόστιμα. Επίκειται άλλωστε ακροματική διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου σχετικά με τον κύριο Σούσκιν, ο οποίος κατηγορείται ότι έχει οργανώσει παράνομες δραστηριότητες, πρόσωπο δηλαδή της αντιπολίτευσης. Επομένως, καταλήγει κανείς το συμπέρασμα ότι οι δυσχέρειες που προκαλούνται στην αντιπολίτευση από το καθεστώς εντείνονται όλο και περισσότερο. Εγώ παρέμεινα ένα διάστημα στη Λευκορωσία και αποκόμισα την εντύπωση ότι η λευκορωσική κοινωνία υποστηρίζει την παροχή οικονομικής βοήθειας, την εκτιμά ιδιαίτερος. Σε ό,τι αφορά τις νέες επενδύσεις θα πρέπει ωστόσο να είναι σαφής η προέλευση των χρημάτων των επενδυωμένων κεφαλαίων και κυρίως τα χρήματα αυτά θα πρέπει να καταλήγουν στις τοπικές αρχές, γιατί αυτές κάνουν καλύτερη χρήση των χρημάτων. Τέλος, θεωρώ ότι οι, οι τελευταίες αποφάσεις έχουν ωστόσο ένα ε, κενό. Είναι δηλαδή άσχημα συντονισμένες. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα επιβάλλουν όρους. Η Λευκορωσία ωστόσο δεν πληρεί τους όρους αυτούς. Μετά έρχονται και λαμβάνουν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί αποφάσεις για τον περιορισμό των κυρώσεων. Από τη δική μου σκοπιά θα ήταν καλύτερο να υπάρχει καλύτερος συσχετισμός χρονικά. Κάτι το οποίο θα οδηγούσε και σε βελτίωση της καταστάσεως στη Λευκορωσία. Εμείς απαιτούμε να βελτιωθεί η εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνια. Αυτό είναι σημαντικό για τους νέους ανθρώπους. Το ίδιο, οι φυτοϊγειονομικοί έλεγχοι στην γεωργία πρέπει επίσης να βελτιωθούν. Το ίδιο δε ισχύει και σε ό,τι αφορά την απελευθέρωση των προξενικών θεωρήσεων. Έρχομαι τώρα στην εκλογική διαδικασία. Και αυτή χρειάζεται σημαντική βελτίωση. Όμως, η λευκορωσική κυβέρνηση δεν κάνει τίποτε προς την κατεύθυνση αυτή. Τον Σεπτέμβριο φέτος θα διεξαχθούν κοινοβουλευτικές εκλογές. Εμείς ενδιαφερόμαστε, ενδιαφερόμαστε πολύ να δούμε την αντιπολίτευση να συμμετέχει. Υπενθυμίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν αναγνωρίζει το Λευκορωσικό Κοινοβούλιο. Πιστεύω όμως ότι πρέπει να γίνει μια προσπάθεια να βελτιωθεί η συνεργασία. Τώρα, κάτι ακόμη. Το μορατόριο μου για την εκτέλεση θανατικών ποινών. Εξακολουθούν ωστόσο να ε, εκτελούνται θανατικές ποινές στη χώρα αυτή. Σε ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές αξίες, το θέμα αυτό για μας έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Τέλος, θέλω να τονίσω ότι εγώ προσωπικά είμαι υπέρ ενός ε, σημαντικά βελτιωμένου ελέγχου των αποφάσεων που έχουν σχέση με τις επενδύσεις στη Λευκορωσία, διότι δεν λέω ότι έχουν γίνει ε, τρομερά πράγματα, αλλά υπάρχουν σφάλματα. Υπήρξαν περιπτώσεις όπου διατέθηκαν κονδύλια χωρίς έλεγχο πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρόκειται για περιορισμένου εύρους ε, σφάλματα, αλλά τα λέω αυτά διότι θέλω να είναι πλήρης η παρέμβασή μου. Εν τέλει, μεν υπέρ των αποφάσεων αυτών, όμως χρειάζεται καλύτερος χρονικός συντονισμός και ε, με τον τρόπο αυτό να αποδώσει και περισσότερα για την υπέρ της Λευκορωσίας. Σας ευχαριστώ για τις διευκρινήσεις. Μας δώσατε βέβαια πολλά επιχειρήματα για μια απάντηση που θα μπορούσε να μην είναι και θετική. Λεωνά Μερεντίν, μπορείτε να μας ε, δώσετε τα φώτα σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Προέρχομαι από την ΓΑΜΑ Δελτανίερ για την ε, Ανατολική Γειτονία. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση αυτή. Να παρευρεθώ εδώ σήμερα το πρωί. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η στιγμή στη διαδικασία των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Λευκορωσία και είναι κάτι που το έχουμε σκεφτεί πολύ προσεκτικά. Θα ήθελα να παρουσιάσω σύντομα κάποιους συναδέλφους που μπορεί να μα βοηθήσουν σε αυτή τη συζήτηση. Ο Καλμάτος που είναι τμήματάρχης από την ΔΕΛΤΑ εκφίν, γιατί η ΕΚΦΙΝ προετοιμάζει τις της πράξης ε, και έχουμε και τον ε, ε, τμήματάρχη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, είναι αρμόδιο για τις εξωτερικές σχέσεις. Αλλά ως διευθυντής από την Κομισιόν, αν μου επιτρέπετε να πω κάποια επεξηγηματικά λόγια και επίσης, αν έχετε και ερωτήσει προ εμένα ή στους συναδέλφου, ευχαριστώ να σας απαντήσω. Καταρχήν, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε μια πολιτική δέσμευση ε, με τη Λευκορωσία ασκώντας ε, κάποια, κάποιο κριτικό πνεύμα. Αυτό ε, είχε να κάνει, όπως σας είπα, με το κριτικό πνεύμα, όμως τα τελευταία ένα-δύο χρόνια μέσω μιας βαθμονομημένης πολιτικής έχουμε καταλήξει σε μια βελτίωση της κατάστασης στη Λευκορωσία. Και μιλάω για μία κάποια βελτίωση, γιατί κανείς δεν ισχυρίζεται ότι η κατάσταση στη Λευκορωσία είναι παρόμοια με αυτή στην Ουκρανία, στην ε, Μολδαβία, αλλά μιλάμε για μια σχετική διαδικασία εδώ. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Υπήρχαν πολλοί άριθμα συμπεράσματα του Συμβουλίου του 2011 και του 2012 που ορθώς είχαν ε, εφαρμόσει αυστηρά μέτρα τα οποία επόπτευε η μαζί με την υπηρεσία εξωτερικής δράσης τα τελευταία 4-5 χρόνια. Ακολουθώντας ε, βάσει της αρχής απόφασης, όπου δεν είχε συμπεριληφθεί η Λευκορωσία στον κατάλογο το 2014, από την περίοδο εκείνη έχουμε δει σαφή αλλαγή στις συνθήκες. Και νομίζω αυτό είναι σημαντικό, γι' αυτό επανερχόμαστε σε εσά και στο Συμβουλίο με μια πρόταση αλλαγή, γιατί πιστεύουμε ότι έχει γίνει ουσιαστική αλλαγή στην κατάσταση. Θα συμφωνήσω με αυτά που είπατε και οι δυο σα για το πόσο σημαντικό είναι αυτό για τους πολίτες της Λευκορωσίας. Εδώ μιλάμε για οικονομικό όφελος και νομίζω ότι όλοι θα συμφωνούσαμε το εξής. Ενώ θα κάνουμε μία παρατήρηση με κριτικό πνεύμα, θέλουμε να δούμε και βελτίωση του επίπεδου ζωής των πολιτών στη Λευκορωσία και αυτό που θέτουμε στο τραπέζι σήμερα αφορά την οικονομική σφαίρα. Και όπως σωστά είπατε, θα μας βοηθούσε να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα που θα βοηθούσε στο να βελτιωθεί η ζωή των πολιτών στη Λευκορωσία. Νομίζω ότι έχουμε ισχυρά κίνητρα να δράσουμε. Τώρα, αν πάμε στον Ιανουάριο του 2015 από το Συμβούλιο έθεσε 29 μέτρα που ήθελε να λάβει η Λευκορωσία. Αυτό ήταν ένα πιθανό βήμα προς τα μπρος, δηλαδή να έρθουμε σε σας με μια πρόταση αν είχαν βελτιωθεί οι προϋποθέσεις και το προκλήθησαμε αυτό εκ του σύνεγγυς. Δεν πρόκειται για μια βιαστική απόφαση λοιπόν που ξαφνικά πήραμε φέτος τον Απριλίο το Μάιο και αποφασίσαμε ότι είναι δραστική αλλαγή. Όχι. Πρόκειται για μια διαδικασία πολύ σταδιακή και πέρσι τον Αύγουστο ήταν μια ζωτική στιγμή όταν απελευθερώθηκαν πολιτικοί κρατούμενοι. Αυτό ήταν ένα βήμα που ελπίζαμε να κάνει Λευκορωσία για πολλά χρόνια. Φυσικά δεν έχει επιλύσει όλα τα προβλήματα, αλλά οδήγησε στις 15 Φεβρουαρίου 2016 στον Άρη Συμβούλιο έναν αριθμό των περιοριστικών μέτρων, όχι όλα τα περιοριστικά μέτρα, κάποια ορθώς τα διατήρησε. Και για μας, για την Κομισιόν και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, αυτό ήταν σημαντικό παράγοντας πυροδότησης, γιατί το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη μας επιβεβαίωσαν με αυτόν τον τρόπο ότι θεωρούσαν και αυτοί ότι υπάρχουν βελτιώσεις όπως υπενθύμησαν στα συμπεράσματα. Και αυτό μας ε, οδήγησε να καλέσουν ο πληρωτής Γενικός Γραμματέας της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης ε, την πρώτη συνάντηση όπου είχαμε έναν ευρύτερο διάλογο με τη Λευκορωσία. Αυτό μας δίνει την ευκαιρία να συζητήσουμε εκ του συνεγγύης πολλά από αυτά τα ζητήματα και φυσικά άκουσα και τις παρατηρήσεις για τη θανατική ποινή, συζητήθηκε το θέμα του μορατόριου στο Μίνσκ νωρίτερα φέτος. Αυτό είναι σημαντικό βήμα Έχουμε δει κάποιες προτάσεις που εκφράζουν ε, τη λύπη τους ακόμη και πρόσφατα. Όμως, το μέτρο που έχουμε εδώ αφορά την οικονομική σφαίρα. Και πιστεύουμε ότι ως τμήμα της ευρύτερη πολιτικής μας ε, στην Ανατολική Γειτονία πιστεύουμε ότι πρέπει να έχουμε πραγματικό αντίκτυπο επιτόπου και για να υπάρχει διαφορά στη ζωή των ανθρώπων, αν θέλουμε να συνεργαστούμε με τους ενωστοτέρους μας στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, πρέπει να έχουμε μεγαλύτερο αντίκτυπο. Εγώ συνάντησα και τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Ε, μεταβήκαμε στη Λευκορωσία μαζί και είχαμε και ειλικρινεί ανταλλαγέ με τους λευκορώσους εταίρους προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι συνθήκες πράγματι πληρούνται, οι προϋποθέσεις πληρούνται πριν να σας παρουσιάσουμε μια τέτοια πρόταση. Πιστεύουμε ότι έχει γίνει σαφής βελτίωση τα τελευταία ένα-δύο χρόνια σε σχέση με το αρχικό έγγραφο που δεν επιλεγόταν Λευκορωσία και βάση και των συμπερασμάτων της 15ης ε, Φεβρουαρίου και της κοινή ε, αποστολή της Κομισιόν και της Ευρωπαϊκής ε, Τράπεζας Επενδύσεων στο Μίνσκ θέσαμε επιτάπητο σε αυτή την πρόταση που πιστεύουμε ότι θα ωφελήσει τους πολίτες της Λευκορωσίας αν μπορούμε να συνεργαστούμε στενότερα στο μέλλον με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Μπορούμε να αναλάβουμε περισσότερες δεσμεύσεις, να εμπλακούμε περισσότερο. Όμως αυτή η πολιτική παραμένει ζωτική, δηλαδή ενίσχυση πολιτική για να σχέση με κριτικό πνεύμα. Φυσικά, είμαστε επικριτικοί, είναι σημαντικός αυτός ο χρόνος, γιατί θα έχουμε και εκλογέ στη Λευκορωσία το φθινόπωρο. Και νομίζω ότι για πρώτη φορά στην Λευκορωσία συμβαίνει και ο διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα στι αρχέ Ιουνίου. Εμεί μαζί με την Υπηρεσία Εξωτερική Δράση παρακολουθούμε από πολύ κοντά την κατάσταση. Και όπω σα είπα, χαίρομαι που είμαι εδώ και ευχαριστώ να απαντήσω σε όποια σχόλια τυχόν έχετε. Ελπίζω να κάλυψα τα κύρια σημεία. Αν θέλετε κάποια άλλη διευκρίνηση, ευχαρίστω. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Keep up, please. Ευχαριστώ. Πολύ λίγα μπορώ να προσθέσω στην πολιτική μας ε, αξιολόγηση που δόθηκε από τον προλήσιδο και από το Στάλφα, από τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑΝΙΑΡ. Ίσως ε, να σας πω ποιο είναι το ιστορικό στο είδος της χρηματοδότησης ε, που κάνουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και η Τράπεζα Επενδύσεων στη Λευκορωσία και σε άλλε χώρε. Ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι ενεργή σε πολλέ χώρε με διάφορα επίπεδα οικονομική ανάπτυξη. Και ακριβώ ε, αυτό είναι το πλαίσιο που λαμβάνει η χώρα αυτή, ε, αυτός ο δανεισμός. Θέλουμε να υποστηρίξουμε οικονομικά και πολιτικά την ανάπτυξη της χώρας και να υποστηρίξουμε τις βελτιώσεις που είδαμε τα τελευταία χρόνια. Όταν πήγαμε στο Μίνσκ, συναντηθήκαμε και με εκπροσώπους άλλων χρηματοοικονομικών οργανισμών, την Παγκόσμια Τράπεζα και την Τράπεζα Νοικοδόμησης και Ανάπτυξης. Ο δανεισμός τους ε, βασικά επικεντρώνεται στον τομέα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και σε κάποιο βαθμό στην τοπική αυτοδίκηση, που ακριβώς είναι οι θεσμοί που μπορούν να υποστηρίξουν περαιτέρω βελτίωση σε πολιτικό επίπεδο στη Λευκορωσία και εμείς θέλουμε αυτός ο δανεισμός ακριβώς να στοχεύσει σε αυτούς τους δικαιούχους και στις τοπικές αρχές και πιστεύουμε ότι αν διευρύνουμε και την εντολή στην Τράπεζα Νοικοδόμησης και Ανάπτυξης θα ευνοήσει αυτό το ωφέλιμο έργο που κάνουν η Παγκοσμία Τράπεζα και η Τράπεζα Γενικοδόμησης και Ανάπτυξης στη Λευκορωσία. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο τώρα στους αδέλφους που θέλουν το λόγο. Κλέρ Μούντι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μετά τα όσα είπε ο συναδελφό μου προηγουμένω, είπατε δηλαδή ότι σημειώνονται κάποιε βελτιώσει στη Λευκορωσία. Αλλά απεκόμισα την εντύπωση ότι υπάρχουν και επιδεινώσεις σε διάφορους τομείς. Άρα λοιπόν πρέπει να εξετάσει κανείς και τις δύο πλευρές του νομίσματος. Δεύτερο, ποιες είναι οι διασφαλίσεις που ισχύουν ήδη. Ναι, είπατε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, κοινωνία, όλα αυτά πρέπει να υποφεληθούν δηλαδή από τις χρηματοδοτήσεις, αλλά πώς θα διασφαλιστούν ότι αυτά δεν θα πάνε σε αυτούς που είναι οι πολιτικοί φορείς στην ε, Λευκορωσία. Και τέλος, ο χρονισμός. Είπατε ότι προβλέπονται εκλογές τον Σεπτέμβριο. Γιατί το εξτάζουμε τα πράγματα αυτά λοιπόν τώρα και όχι αργότερα μέσα στο έτος. Δεν έχει μικρό, μικρόφωνο ο πρόεδρος, δυστυχώς δεν έχει μικρόφωνο. Εσείς κύριε, εσείς κύριε Στρογεύσκη. Θα ακολουθήσει ο κύριος Κέρμελ. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας. Είχα την πρόθεση να σας επισημάνω ότι είναι αναγκαίο οι αποφάσεις και η εκτέλεση των αποφάσεων για τη Λευκορωσία να συντονιστούν καλύτερα. Το σημείο κλειδί είναι οι εκλογές του Σεπτεμβρίου. Εδώ πρέπει να επιβληθούν όροι. Δηλαδή πρώτα συμμετοχή όσων επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εκλογές. Εκεί έχουμε ένα σημαντικό πρόβλημα. Δεύτερο, η ίδια η προεκλογική διαδικασία. Πρόσβαση ιδίω στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εκεί παίζει ένα σημαντικό ρόλο ο ίδιος ο Λουκασένκο. Σε ό,τι αφορά τους αποδέκτες της, ε, των ενισχύσεων, εκεί όπου τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε τοπικές αρχές, σε μικρές και μέσες επιχειρήσεις, εκεί η αποτελεσματικότητα των ελέγχων πρέπει να είναι εγγυημένη. Όμως οι δαπάνες στην διοίκηση, τις οποίες θα κάνει η ίδια η κυβέρνηση, εκεί πολλοί έχουν επιφυλάξεις σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις από πλευράς Ευρώπης και για τα σχέδια τα οποία χρηματοδοτήθηκαν τα τελευταία 5 έως 7 χρόνια. Υπήρξε πρόοδος. Ναι, υπήρξε πρόοδος. Η πρόοδος αυτή ήταν ικανοποιητική. Δυστυχώς όχι. Γι' αυτό και οφείλουμε να ασκήσουμε εντονότερη πίεση ώστε τα πράγματα αυτά να υλοποιούνται στον προβλεπόμενο χρόνο. ώστε να ωφελούνται πραγματικά οι δικαιούχοι των ε, στηρίξεων. Άρα χρειάζεται πολύ καλύτερος σχεδιασμός και μεγαλύτερη πίεση. Είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη αυτά. Ευχαριστώ. Εσείς κύριε Κέρμελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και όλους τους προλαλήσαντες. Επιθυμώ να συμφωνήσω με την κυρία Μούντι ιδίω. Θεωρώ ότι στο πλαίσιο αυτό πρέπει να στήσουμε ένα πολύ καλό monitoring. Για παράδειγμα ένα κατάλογο στον οποίο θα περιλάβουμε τα προβλήματα που διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν. Πάντοτε θα υπάρχει ένα θέμα ερμηνεία, εάν δηλαδή τα όσα επιτεύχθηκαν αποτελούν πρόοδο ή όχι. Αλλά θα πρέπει να σημειωθούν τα προβλήματα που υπάρχουν και ιδίω ποιου στόχους έχουμε. Διότι αλλιώ φοβούμε σε ένα-δύο χρόνια, όταν θα στρέφουμε τα βλέμματα προς τα πίσω, δεν θα μπορούμε τελικώς να κρίνουμε αν οι προσπάθειές μας απέβησαν επιτυχής ή όχι. Γι' αυτό νομίζω πρέπει ε, να ξεκαθαρίσουμε πού εντοπίζονται τα προβλήματα, τι θέλουμε να επιτύχουμε, ώστε να έχουμε στο προσεχές μέλλον συγκεκριμένες παραμέτρους για να μπορούμε να μετρήσουμε την ε, πρόοδο που θα έχει ενδεχομένω επιτελεστεί. Άλλος... Δεν Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι ο Ντεκ Σούμπολ από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Νομίζω ότι ακούσατε από τον συνάδελφο είμαι. Νομίζω ότι θα μπορέσω ενδεχομένως να απαντήσω σε κάποια από τα σημεία που έθιξαν τα μέλη της Επιτροπής. Καταρχήν, ναι, υπάρχει σημαντική πρόοδος από την αρχή του 2014 και αυτό από τη στιγμή που απελευθερώθηκαν οι πολιτικοί κρατούμενοι. Έχουμε όμως και κάποια άλλα ενθαρρυντικά σήματα, περισσότερη συμμετοχή της Λευκορωσίας ε, στην σύμπραξη, καλύτερη συνεργασία, το θέμα της απελευθέρωσης των θεωρήσεων, αλλά και το θέμα της εταιρική σχέσης για καλύτερη κινητικότητα. Βεβαίως υπάρχουν ακόμα κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες δεν έχουν αποσαφινιστεί, αλλά το σημείο το πιο σημαντικό είναι η εργασία που γίνεται στα πλαίσια της ομάδας συντονισμού. Εκεί τους κάνουμε κάποιες παρουσιάσεις για το ευρωπαϊκό κεκτημένο κάτι που δεν γνωρίζουν και βεβαίως συνεχίζει η ενημέρωση, είναι η πρώτη φορά που συναντηθήκαμε επί μια μισή μέρα με φορείς της κοινωνίας των πολιτών, με εκπροσώπους των ε, διαφόρων οργανώσεων και νομίζω ότι η δεύτερη σειρά συζητήσεων που θα λάβει η χώρα θα είναι ακόμα πιο επικοδομητική. Η συμφωνία του Μίνσκ, όπως ξέρετε, έχει λάβει χώρα στην ε, Λευκορωσία. Δεν ήταν εύκολο να αποφασιστεί ο χώρος, ο τόπος στον οποίο θα γίνουν αυτές οι συζητήσεις διαπραγματεύσεις, ιδιαίτερα από μέρους της Ρωσίας. Τελικά όμως βλέπουμε ότι ο ρόλος που έπαιξαν ήταν πολύ επικοδομητικός. Άκουσα πολύ προσεκτικά τον ε, εκπρόσωπο της ε, Λευκορωσίας και βεβαίως και εμείς ανησυχούμε όσον αφορά από τα σημεία που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, την θανατική ποινή. Συμμετείχατε εξάλλου και εσείς ε, στην συζήτηση που έλεγε χώρα για την νομοθεσία καθώς και τις κοινοβουλευτικές ε, εκλογές του Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα να πω ότι σε κάθε περίπτωση βλέπουμε πρωτοβουλίες από μέρους της ε, Λευκορωσίας για θέματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Λευκορωσία θέλει να συμμετάσχει στον ε, διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό θα συνεχιστεί στις 7 Ιουνίου στο Μίνσκ με συμμετοχή από μέρους Ευρωπαϊκής Ένωσης του επικεφαλής της υπηρεσίας μας. Ο κύριος Λαμπρινίδης, Επιτρόπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, θα είναι επίσης παρόν και μάλιστα είχε και μια συνάντηση δυόμιση ωρών με τον πρόεδρο Λουκασέγκο και συζητήθηκαν θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και η θανατική ποινή. Οργανώνεται μάλιστα και μία συνδιάσκεψη με θέμα την θανατική ποινή ε, με συμμετοχή και πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ε, είδατε μάλιστα ότι ο πρόεδρος Λουκασέγκο συναντήθηκε και με τον Πάπα στη Ρώμη και μάλιστα ζητήθηκε από τον κύριο Λουκασέγκο από μέρους του Πάπα Φραγκίσκου να γίνει κάτι σε σχέση με την κατάργηση της θανατικής ε, ποινής. Η αντίδρασή του δεν ήταν αρνητική. Οργανώνεται λοιπόν από κοινού με την Επιτροπή της Βενετίας ε, του Συμβουλίου της Ευρώπης η συνδιάσκεψη για την θανατική ποινή και βεβαίως θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης δικαστών, συμμετοχή των γυναικών ε, στην πολιτική και ανθρώπινα δικαιώματα. Όλα αυτά τα θέματα τα επεξεργαζόμαστε από κοινό με το Συμβουλίο της Ευρώπης με κάποια απτά αποτελέσματα, αν και πολλά ακόμα πρέπει να γίνουν. Πρέπει να πούμε ότι η διαδικασία έχει αρχίσει να κινείται. Η Λευκορωσία λοιπόν έχει ξεκινήσει προς την κατεύθυνση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και βεβαίως ελπίζουμε ότι θα συνεχίσει την πορεία της προς αυτή την κατεύθυνση. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ και στις εκλογές που θα λάβουν χώρα στις 11 Σεπτεμβρίου, κοινοβουλευτικές εκλογές και βεβαίως υπάρχει και η εναλλακτική να αναβληθούν οι εκλογές, να καθυστερήσουν ή να συζητηθεί το θέμα λίγο νωρίτερα. Βεβαίως ξέρουμε ότι υπάρχει η προεκλογική εκστρατεία, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία. Ελπίζουμε να βελτιωθεί σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές. Κάτι που βεβαίως θα δικαιολογήσουν και τις πρόσφατες κινήσεις μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ για τις διευκρινήσεις σας. Καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολη η θέση μας. Οι εκπρόσωποι της Επιτροπής είναι πολύ σήμερα εδώ. Παρ' όλα αυτά τα μέλη της Επιτροπής μας απουσιάζουν. Τα θέματα είναι πολύ σημαντικά. Οι διερμηνείς θα διακόψουν γιατί ήδη έχουν ξεπεράσει το κανονικό του ωράριο και του ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν πολλοί αστάθμητοι παράγοντες. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν μπορεί να κάνει κάτι. Όσον αφορά το δημοσιονομικό κομμάτι αυτής της επιχείρησης, εάν προχωρήσει σε δανεισμό η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χωρίς τις εγγυήσεις των, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αυτοί που θα πρέπει τελικά να χρηματοδοτήσουν θα είναι τα κράτη-μέλη. Αν υπάρξει εγγύηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεσμεύεται ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ λοιπόν ζητούμε περαιτέρω κονδύλια για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η θέση μας είναι δύσκολη. Δεν υπάρχει πρόβλημα νομίζω να δανείσει κατευθείαν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στην Λευκορωσία. Έτσι δεν είναι και εδώ απευθύνομαι στον εκπρόσωπο της ΕΚΦΙΝ. Υπάρχει πρόβλημα στο να δανείσει κατευθείαν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στη Λευκορωσία. Στην θεωρία όχι. Στην πράξη όμως υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει συμφωνία πλαίσιο καταρχήν μεταξύ της τράπεζας και της Λευκορωσίας και ενδεχομένως δεν ε, θα υπογραφεί μια τέτοια συμφωνία πλαίσιων εάν δεν τροποποιηθεί η συμφωνία. Υπάρχει επίσης η δυσκολία να δανείσει η τράπεζα εάν δεν υπάρχουν αυτές οι εγγύησει. Χωρίς την εγγύηση δηλαδή του, του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενδεχομένως μπορεί να υπάρξει δανεισμός στα πλαίσια του σημερινού ποσού, χωρίς δηλαδή επέκταση του ε, ποσού. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Υπάρχουν τόσο λίγα μέλη της Επιτροπής μας στην αίθουσα που νομίζω ότι οφείλουμε να ολοκληρώσουμε. Εχθές, στη διάρκεια της συνεδρίασής μας, και στη διάρκεια της συνάντησης των συντονιστών αποφασίζαμε να διοριστεί η κυρία Κάλιο Σαμπάλ σαν εισηγήτρια. Εάν αρνηθεί αυτόν το ρόλο, θα το αναλάβω εγώ. Σας προτείνω λοιπόν να μου αναθέσετε τις επαφές με την πιθανή εισηγήτρια και να αποφασίσουμε αν ναι ή όχι θα υποβάλουμε έτοιμα για αντίθεση, αντίρρηση. Yes. Uh, if I may, President, uh, just uh, uh one, uh, a couple of additional words from, from my side uh, on this specific point of